Uh, Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Ας αρχίσουμε. Αλλά ο κύριος, ο συνάδελφος που είναι υπεύθυνο για το πρώτο θέμα θα έχει καθυστέρηση. Ο κύριος Μπιζόη. Δεν θέλω όμως να αφήσουμε πολύ μεγάλο κενό. Είμαστε αρκετοί εδώ. Ο Γούλφερ εκπροσωπείται, οπότε μπορούμε κάπως να θέσουμε κάποια θέματα. Εν πάση περιπτώσει, πρώτον, καλωσορίσατε σε αυτή τη διήμερη συνεδρίαση, θα γίνει σήμερα και αύριο. Καλωσορίσετε, θέλω να καλωσορίσω και το ακροατήριο που μας ακούει μέσω του διαδικτύου. Θα ακούσετε, θα έχετε την τελευταία προσθήκη των ειδήσεων, αλλά βεβαίως αυτό έχει ανεβεί και στην ιστοσελίδα μας και επίσης μπορείτε να ενταχθείτε στους φίλους της Επιτροπής και να παίρνετε το κείμενο αυτό κάθε μήνα και να έχετε άμεση πρόσβαση στα έγγραφα. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για όσους είστε φίλοι της ενιαίας αγοράς. Θέλω λοιπόν να σας ζητήσω να εγκρίνουμε και επισήμως την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης αυτής, η οποία είναι αρκετά φορτωμένη. Υπάρχουν πολλά θέματα για τα οποία θέλουμε τροπολογίες και αύριο θα γίνουν και ψηφοφορίες. Θα εξετάσουμε αύριο τις ε, τροπολογίες του πακέτου της κυρίας Ρότεμπερκ και θα γίνουν και ψηφοφορία. Η μόνη διαφορά είναι ότι η γνωμοδότηση του κυρίου Χασκόψκη έχει αφαιρεθεί από την ημερήσια διάταξη, γιατί δεν έχουμε τις τροπολογίες σε όλες τις ε, γλώσσες. Γι' αυτό μου είπαν ότι θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε και να ψηφίσουμε στις 17 Σεπτεμβρίου. Ο κύριος Τρασκόφσκι λοιπόν δεν θα συμπεριληφθεί στη σημερινή ημερήσια διάταξη. Και ίσως να, να χρησιμοποιήσουμε έτσι κι αλλιώς ε, την μισή ώρα που θα δίναμε σε αυτή την έκθεση γιατί είναι φορτωμένη. Λοιπόν, έγκριση της Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω να ανακοινώσω σε όλους και στο διαδίκτυο, τους ακροατές του διαδικτύου, ότι ο κύριος Σιλικιώτης, ο οποίος εδώ με βοηθάνε για να λέω σωστά τα ελληνικά ονόματα, λέει ο Πρόεδρο. Ο κύριο Σιλικιώτη, λοιπόν, υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανία, Τουρισμού και Ανταγωνιστικότητα της Κύπρου και ο οποίο θα προεδρεύσει το Συμβουλίο Ανταγωνιστικότητα κατά τη διάρκεια τη Κυπριακή Προεδρία, θα έρθει στι 3 αύριο το απόγευμα στην Επιτροπή μα. Ελπίζω ότι πολλά μέλη θα παρευρεθούν. Επίσης, οι συντονιστές έχουν προσκληθεί να φάμε όλοι μαζί μαζί του. Αύριο ε, έχουμε ένα ιδιαίτερο μεσημεριανό ε, γεύμα για εκείνον πριν ε, έρθει να απευθυνθεί στην Επιτροπή μας. Κάποιοι από μας. Είχαμε πάει σε αποστολή στην Κύπρο, τον έχουμε συναντήσει και ξέρω ότι είναι εξαιρετικά ενθουσιώδης για τις εργασίες της Επιτροπής μας. Και κατά τη συνεδρίαση εκεί συναντηθήκαμε με τους πρόεδρους των πέντε ομάδων εργασίας ε, των βασικών μας θεμάτων μας, συμπεριλαμβανομένων και των ε, δημοσίων συμβάσεων η Κύπρος είναι πολύ προηγμένη στο θέμα των δημοσίων προμηθειών, κυρίως των ηλεκτρονικών προμηθειών. Έχει γίνει την περασμένη εβδομάδα, ή μάλλον πριν δύο εβδομάδες, ένα ειδικό σεμινάριο στο Κοινοβούλιο γι' αυτό, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας παρακαλώ λοιπόν αύριο στις 3 το απόγευμα να έρθετε εδώ. Επίσης θα ψηφίσουμε το πακέτο της κυρίας Ρόιτεμπερκ στην Τρίτη το απόγευμα. Θα έχουμε δύο χρόνους ψηφοφοριών αυτή την εβδομάδα. Ο ένας 10 στις 12 και ο άλλος από τις 45 μετά το κλείσιμο αυτής του θέματος και τις ομιλίες του κυρίου Σικιώτη. Όπως ήδη σας είπα, θα αναμεταδίδεται ζωντανά μέσω διαδικτύου συνεδρίαση αυτή και υπάρχει και ένα μήνυμα προς εσάς από τις 7 Ιουνίου. Έχουμε τα πρακτικά τα οποία θα έχουν εγκριθεί μέχρι το τέλος της συνεδρίας Επιτροπής αν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις. Περιμένουμε τον κύριο Μπουζόη που είναι ο για το πρώτο θέμα. Θέλω όμως να επισύρω την προσοχή σας και αν θέλει κάποιος να σχολιάσει, πολύ ευχαρίστως. Θα έχετε δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28 και 29 Ιουνίου, που ήταν το τελικό συμβούλιο κατά την Προεδρία της Δανίας. Θα έρθει, ήρθε και ο, πρόεδρος, ε, ο Υπουργός Χολιζών. Θα θυμόσαστε ότι στο ψήφισμά μας ως Επιτροπή για το πακέτο της ενίας αγοράς που μας παρουσίασε ο κύριος Μπαρνιέ τον Ιούνιο. Αναφέραμε συγκεκριμένα ότι θέλαμε να βελτιωθεί η διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς και θεωρούσαμε συγκεκριμένα ότι υπάρχουν τομείς όπου επιδόσει των κρατών μελών στην εφαρμογή και την επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς όπως επίσης και της παρακολούθησης και των επιδόσεων θα πρέπει να ελεγχθούν έτσι περαιτέρω στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι στα συμπεράσματα του Συμβουλίου οι Πρωθυπουργοί ρητά αναφέρουν και σας διαβάζω. Τα κράτη-μέλη και η Επιτροπή θα εξασφαλίσουν την καλύτερη εφαρμογή και επιβολή των κανόνων της Ινέας αγοράς και η Επιτροπή θα παρακολουθήσει τις επιδόσεις επιλαμβανομένης μιας ετήσιας έκθεσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ ευτυχείς εμείς που ήδη το έχουμε υποστηρίξει αυτό σαφέστατα. Το επισήμανα στην διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών, γιατί θα χρειαστούν κάποιες επιτροπές στον τρόπο οργάνωση των Επιτροπών σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, γιατί αυτή τη στιγμή η Επιτροπή Απασχόλησης και η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων είναι οι αρμόδιες για, τα, για τις εκθέσεις των ε, εξαμήνων για τα οικονομικά θέματα. Εδώ όμως πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί εμείς. Πρέπει να γνωρίζετε ότι τα κράτη-μέλη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δηλαδή, συμφώνησαν με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες επί της οποίας θα κάνουμε έκθεση και λέει ότι είναι ευπρόσδεκτη αυτή η ανακοίνωση και πρέπει άμεσα να υλοποιηθεί συμπεριλαμβανομένης και μια ταχείας δράσης για την αφαίρεση των αδικαιολόγητων εμποδίων. Επίσης συμφώνησαν με την ανακοίνωση για την διακυβέρνηση της ε, ενιαίας αγοράς. Θα γίνουν και αυτές εκθέσεις ε, ιδίας πρωτοβουλίας. Είναι σοβαρή δουλειά αυτή που θα κάνει η Επιτροπή μας μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Θέλω λοιπόν να επιστήσω την προσοχή σας στις επιπτώσεις του ψηφίσματος που κάναμε για την ενιαία αγορά. Άλλα σχόλια υπάρχουν. Ο κύριος Σβάμπα. Ευχαριστώ για αυτή την παρουσίαση της δουλειάς μας σε σχέση με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε. Σωστά είπατε ότι και οι δύο επιτροπές, η ΕΚΟΝ και η ΕΜΠΛ, αυτή τη στιγμή ασχολούνται με το ε, περιεχόμενο του Ευρωπαϊκού ε, Εξαμήνου και δεδομένου ότι εμείς όλοι, ειδικότερα όταν ε, Θέλουμε να μιλήσουμε για την τελευταία αποφάσει των συντονιστών ότι αυτό το θέμα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην εσωτερική αγορά. Ε, σημαίνει αυτό ότι πρέπει να βρούμε μια τεχνική λύση για να μπορέσουμε να έχουμε μια επαρκή συμμετοχή σε αυτό το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Ευχαριστώ. Έχω αρχίσει να εργάζομαι από αυτό. και ενδεχομένως να είναι και υπόθεση δύναμης το Συμβούλιο είπε στο πλαίσιο των συζητήσεων ε, του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και όχι στις υφιστάμενες συζητήσεις. Έτσι λοιπόν ίσως να υπάρχει μια, μια παράλληλη οδός που να μας ταιριάζει καλύτερα για να εμπλέκονται όλες οι επιτροπές που ασχολούνται όπως και εμείς με την έννοια αγορά, μεταφορές, ενέργεια κτλ. Και ξέρω ότι οι συνάδελφοι σε αυτά τα θέματα, κυρίως ο κύριος Σίμψον, το γνωρίζετε πολύ από εσά, ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να υπερασπιστεί μια ισχυρότερη έγκριση, θέσπιση των κανόνων της ενιαίας αγοράς στον τομέα των μεταφορών και ιδίω των σιδηροδρόμων. Κύριε Γκέφαρτ. Ε, Ευχαριστώ και εγώ στους ίδιους τόνους να πω ότι με εξέπληξε που η Επιτροπή ΙΜΚΟ δεν είχε ε, συμμετάσχει σε ίσους όρους ε, και ίσως θα ήταν καλύτερο να έχουμε ένα πλαίσιο, ίσως παράλληλα, ώστε να επηρεάσουμε κι εμείς ε, τις διαδικασίες, ε, γιατί η εσωτερική αγορά είναι η ουσία της εξέλιξης και πρέπει να σας ζητήσω, κύριε Πρόεδρε, ως πρόεδρο αυτής της Επιτροπής ε, στεναρά να συμμετάσχουμε σε αυτήν την, την συζήτηση. Πραγματικά με εξέπληξε η απόφαση των ε, Προέδρων του Κοινοβουλίου. Δεν είχα ενημερωθεί εκ των προτέρων ότι προετοιμαζόταν κάτι τέτοιο και αυτό πραγματικά δεν είναι σωστό. Η εσωτερική αγορά δεν είναι κάτι κάπου στο περιθώριο. Είναι ε, στο κέντρο αυτού του ζητήματος και η Επιτροπή μας είναι οριζόντια Επιτροπή. Όταν δεν είναι ΙΜΚΟ, λοιπόν, ε, ποιο ε, είναι υπεύθυνο και αρμόδιος ε, η Επιτροπή Μεταφορών, εντάξει, είναι και αυτή, αλλά εμεί είμαστε μια οριζόντια Επιτροπή και γι' αυτό είμαστε πολύ σημαντικοί. Όπως σας είπα, αυτό το οποίο θα συμβεί και αυτό που επιδιώκουμε είναι να έχουμε μια δική μας κατεύθυνση, κυρίως για την αγορά. Και είμαι βέβαιος ότι αυτό θα το στηρίξετε κι εσείς. Άλλοι συνάδελφοι. Right, okay. um, in which case... Οπότε, ο κύριος Μπουσόη δεν είναι Οι σκιώδεις θέλουν να ξεκινήσουν ή μήπως βρίσκεται εδώ ε, η κυρία Μακλάρκιν για το επόμενο θέμα. Γιατί έτσι κι αλλιώς θα ήταν πολύ σύντομη ανταλλαγή απόψεων γιατί. Ε, για το θέμα του κυρίου Μπουζόη. Μήπως να ε, συμφωνείτε οι να ξεκινήσουμε με την κυρία Μακλάρκιν. Για... Ε, Είμαστε λίγο νωρίτερα με την έκθεση της κυρίας Μακλάρκιν, πρόγραμμα για την αντιγανιστικότητα των επιχειρήσεων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Δεν βρίσκεται εδώ ο κύριος Σμιτ, ο κύριος Κρότσμαν, δεν ξέρω. Μπορεί να τον αντικαταστήσει η κυρία Ρούλε. Η Επιτροπή βρίσκεται εδώ για τα θέματα των μικρομεσαίων. Περιμένουμε την κυρία Φραντσέσκα. Όχι, κάποιον άλλον περιμένουμε από την Επιτροπή. Εν πάση περιπτώσει, η Επιτροπή βρίσκεται εδώ. Οπότε, κυρία Μακλάρκιν, αν δεν έχετε αντίρρηση, ας ε, ασχοληθούμε με τις ε, τροπολογίες αυτές μετά θα σχολιάσουν οι σκιώδεις. Κυρία Μακλάρκιν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Πολύ σπάνια είμαι τόσο νωρίς για οτιδήποτε και αυτό καταδεικνύει ότι με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα αυτά τα θέματα γιατί μιλάμε για την ανταγωνιστικότητα για τις μικρομεσαίες. Κάτι το οποίο με απασχολεί, με έχει απασχολήσει ιδιαίτερα. Μιλάμε για βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά των ΜΜΕ. Αυτό το υποστηρίζω ιδιαίτερα και θα βρείτε και αρκετές τροπολογίες που ενισχύουν αυτή την ιδέα. Επίσης, ε, έθεσα τις ΜΜΕ στο επίκεντρο και έκρινα ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει μεγάλος φόρτος. Επίσης να έχουμε ευφυείς κανονισμούς και να απλουστεύουμε το πλαίσιο λειτουργίας. Και όταν αντιμετωπίζουμε κρίση να μπορούμε να τις βάλουμε στο επίκεντρο των μελημάτων μας. Δεν θα πρέπει να γίνονται επικαλύψεις στο έργο των κρατών μελών, γι' αυτό θα πρέπει μέσα τα πλαίσια του ευρωδικτύου Ευρωπαϊκού Δικτύου με τις ΜΜΕ να είμαστε σίγουροι ότι οι τράπεζες μπορούν να προβάλλουν όλες τις εγγυήσεις υπέρ των ΜΜΕ και να παρουσιάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα εκθέσεις ανάπτυξης. Με τους σκιώδους, με συγχωρείτε, συναντηθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα και φτάσαμε σε σαφείς συμβιβασμούς έτσι ώστε να προβάλλουμε τα spin-offs και τη δεύτερη ευκαιρία για τις ΜΜΕ, έτσι ώστε να, μπορέσουμε να, να μπορέσουν να συνεισφέρουν και στο ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, τονίσαμε τη σημασία του δικτύου αυτού και στο θέμα του τουρισμού φτάσαμε σε ε, σε, συγκεκριμένα, σε συγκεκριμένες προτάσεις συμβιβασμού και χαίρομαι γιατί όλες οι ομάδες υποστήριξαν αυτούς τους συμβιβασμούς. Γι' αυτό προτείνω κάπως έτσι να διατυπωθεί και η τροπολογία 9. Ελπίζω να την υποστηρίξετε γιατί ε, μοιάζει με τις 6 και 7 του κυρίου Σμιτ και θα ήθελα να κρατήσουμε και την 12. Ε, επίσης, μερικές καταπίπτουν του κυρίου Σμιτ και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να φτάσουμε σε, σε ένα συμβεβασμό στον κατάλογο ψηφοφοριών. Η ε, γραμματεία θα βρει την καλύτερη εκδοχή. Ελπίζω οι τροπολογίες μου να γίνουν αποδεκτές, ιδιαίτερα σε σχέση με ε, απονομή βραβείων και επάθλων. Δεν θα πρέπει να είναι μια δαπανηρή διαδικασία και πιστεύω ε, και χαίρομαι που είναι εδώ ο κύριος Κρόιτσμαν και ελπίζω στην Επιτροπή Ήτρε να προωθήσει την άποψή μας. Αύριο το πρωί θα ψηφίσουμε και θα ήθελα να συζητήσουμε εκτενώς την πρόταση σήμερα το απόγευμα για να έχω την υποστήριξή σας αύριο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Όλα τα μέλη έχουν τον κατάλογο όλων των τροπολογιών συμβιβασμού. Στα αγγλικά οπωσδήποτε. Ας δούμε ποια είναι η άποψη των σκιωδών. Ο κύριος Μπαλτασάρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκτιμήσαμε ιδιαίτερα την εργασία της εισηγήτριας που προσπάθησε να συμβιλιώσει όλες τις απαιτήσει υπό το φως του βασικού στόχου, δηλαδή της αρρωγής προς τις ΜΜΕ, έτσι ώστε να υπάρχει ένα νέο συμμετοχικό σχήμα εκτιμήσαμε τη θέλησή της να ελαφρυνθεί ο γραφειοκρατικός φόρτος που επιβαρύνει τις ΜΜΕ με μία σειρά κανόνων και κανονισμών, δηλαδή ενός επιβαρημένου ρυθμιστικού πλαισίου. Θεωρούμε ότι το θέμα τραπεζικής της τραπεζικής εποπτείας προσκρούει σε δυσκολίες μέσα στα πλαίσια αυτής της αρρωγής και των εγκυοδοτήσεων καθώς και της ε, δανειοληψίας των ΜΜΕ. Και δυστυχώς το τραπεζικό σύστημα δίνει πολύ λίγες απαντήσεις, πολύ περιορισμένες. Γι' αυτό θα πρέπει να εποπτεύουμε καλύτερα τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος Εκτιμήσαμε στο, το γεγονός ότι αναφέρεται στις μικροεπιχειρήσεις, δηλαδή στις βιοτεχνίες περισσότερο, λαμβάνοντας υπόψη ένα το ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, χωρίς να μιλήσουμε για προτιμήσεις. Συμφωνούμε με τις ε, τροπολογίες συμβιβασμού, προτείναμε αυτό λοιπόν το στόχο, ως προς το παράρτημα 1 υπάρχουν διαφοροποίησεις. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να μιλήσουμε για τη νέα αρμοδιότητα της Επιτροπής σε θέματα τουρισμού. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν μιλάμε για το περιεχόμενο του προγράμματος COSME. Ε, είμαστε ικανοποιημένοι από την έκβαση της εργασίας γενικά. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Μακλάρκιν για την αποφασιστικότητά της και για την ε, παραγωγική συνεργασία μας. Είμαι ιδιαίτερος ικανοποιημένος που η γνωμοδότηση αυτή αναφέρεται σε επιχειρηματίες που προέρχονται από μεταναστευτικές, από οικογένειες μεταναστών και που έχουν την ευκαιρία να τους δοθεί η δεύτερη αυτή ευκαιρία. Μια δεύτερη ευκαιρία είναι καλό να, να προωθούμε την αλλαγή γενεάς στις επιχειρήσεις. Πιστεύω ότι αυτή η γρομοδότηση θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε τους στόχους της στρατηγική της Ευρώπης 2020 για να προωθήσουμε τη θέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι πραγματικά ο κινητήρας της οικονομικής μας ανάπτυξης. Υπό την έννοια αυτή, είναι βασική η θέση του στην προσπάθειά μας να αναπτύξουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εξάλληψη της ανεργίας των νέων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ρέπολ. Ο κύριος Κρότσμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω καταρχήν να πω δύο λόγια εκ μέρους του συναδέλφου Όλη Σμιτ που δεν μπορεί να παρευρεθεί και λέει στο έγγραφο που μου έδωσε ευχαριστούμε την εισηγήτρια για το έργο των συμβιβαστικών τροπολογιών. Συμφωνούμε ότι δεν θα πρέπει να Θα πρέπει να φροντίζουμε ότι όλοι θα έχουν σαφείς πληροφορίες. Πρέπει να στηρίξουμε τις στοχευμένες πληροφορίες για τους νέους και ε, νέους επιχειρηματίες συμφωνεί με την εισηγήτρια ότι το στο πρόγραμμα πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι. Χαίρεται που περιλαμβάνεται και η δεύτερη ευκαιρία για τους επιχειρηματίες. Αυτό ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές είναι οι λίγες προτάσεις που μου έδωσε στο κείμενό του. Θέλω να πω και εγώ δύο λόγια γιατί είμαι εισηγητή επί του θέματος στην Επιτροπή Ήτρα. Όπως ε, είπε και ο κ. Μπαλταζάρ, κ. Ραντζάν, ενδιαφέρεται να συμπεριληφθεί ο τομέας του τουρισμού και γνωρίζουμε ότι και οι Ιταλοί και οι Ισπανοί φίλοι ε, συμφωνούν. Εγώ, κύριε Παλτασάρη, το είπα ειλικρινά, δεν τον βρίσκω αυτό, ε, δεν βρίσκω αυτό να έχει νόημα, γιατί δεν αναφέρεται κανένας τομέας. Θα πρέπει βεβαίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτού του κλάδου να αναφέρονται όταν χρειάζεται. Εγώ ε, το αφαίρεσα, αφαίρεσα την αναφορά ε, εξακολουθεί να αναφέρεται βέβαια στην τροπολογία, αλλά για μένα αυτό δεν έχει νόημα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Στη... Προσπάθησα να πετύχουμε τρία βασικά πράγματα. Πρώτον, η μείωση της γραφειοκρατίας είναι πολύ σημαντική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεύτερον, η βελτιωμένη πρόσβαση στις αγορές και η καλύτερη ε, πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Αυτή είναι η βασική στόχη βεβαίως. Μπορείτε να με υποστηρίξετε στον προϋπολογισμό. Γνωρίζετε ότι η Κομισιόν δίνει 2,5 μόνο δισεκατομμύρια ευρώ γι' αυτό. Αν δούμε όμως τον ορίζοντα 2020 υπάρχει το 15% σχεδόν είναι ο συνολικός προπολογισμός του 2020 φτάνουμε στα 8-9 δισεκατομμύρια ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι καλό να διπλασιαστεί το ποσό, όχι βεβαίως να φτάσουμε τα 9 δισεκατομμύρια όπως τον ορίζοντα 2020, αλλά κάθε επιχείρηση, κάθε μικρομεσαία επιχείρηση που καινοτομεί θα πρέπει να πάει στο πρόγραμμα του ε, ορίζοντα 2020 και όλα τα άλλα να μείνουν εδώ. Αυτό σημαίνει ότι ίσως όταν ε, το προσπαθήσουμε αυτό μπορούμε να διπλασιάσουμε τον προϋπολογισμό και να έχουμε περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα αλλά έμαθα ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσω αυτής της έκθεσης. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Καταρχήν, αν, ανέφερα τον ορίζοντα 2020, αλλά αυτό είναι ε, άλλο θέμα. Οι αρμόδιοι όμως για τον ορίζοντα 2020 δεν έχουν πρόβλημα με αυτό. Αυτά είναι τα θέματα που θέλω να αναφέρω πέρα από αυτά που ε, μου έγραψε ο συνάδελφος και σας διάβασε. Ευχαριστώ. Thank you very much. of course, within the... Ευχαριστώ. Στην Επιτροπή ε, δι... όπου ασχολείστε με τον ορίζοντα 2020 θα μπορέσετε την πρόταση αυτή να την υποβάλλετε. Κυρία Ρούλα. Και εγώ συμφωνώ με τους σκιώδες στην Ήτρε ε, που θα υποστηρίξουν έτσι λοιπόν και εγώ σας υποστηρίζω πλήρως. Ε, ε, υπάρχουν και κάποια σημεία στα οποία είμαι λίγο... Ε, ας πούμε, επιφυλακτική. Τι είναι το red tape, είναι η γραφειοκρατία. Αυτό θα ήταν σωστό, αλλά συνήθως όταν μιλάμε για red tape, μιλάμε για υπερβολική ρύθμιση. Ε, όντως χρειαζόμαστε λιγότερη ρύθμιση, αλλά πού. Εγώ έκανα μια μελέτη για την δημιουργία μηχανών στο Ιμβάντι Βιντεμβέργη και εκεί φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κάτι τέτοιο, γιατί ανοίγει τις αγορές, ε, νέες αγορές και δεν είναι νέα κίνητρα. Έτσι λοιπόν ζητώ λίγο να ε, προχωρήσουμε αυτό το θέμα της συζήτησης της υπερβολικής ρύθμισης και να δούμε τι ακριβώς εννοούμε με αυτό. Αν είναι ε, η γραφειοκρατία Εντάξει, αλλά αν είναι ε, συγκεκριμένες νομοθεσίες που πάνε προς ε, την κατεύθυνση της καινοτομία, θεωρώ ότι αυτές ε, δεν είναι υπερβολική ρύθμιση, είναι απαραίτητες και γι' αυτό θα ζητούσα να μην υπάρχει εκεί συμβιβασμό. Επίσης, αυτό που αναφέρεται για τον τουρισμό το θεωρώ σωστό και θα συμφωνήσω με την κυρία Μιτλάρκιν, γιατί ο τουρισμός είναι ε, κάτι με το οποίο κανείς, χωρίς το οποίο κανείς δεν μπορεί να ζήσει και εγώ το προτιμώ και θέλω να βρίσκεται εκεί μέσα στην έκθεση. Ευχαριστώ. Good. Um, any other members? Άλλο μέλος που θα ήθελε να πάρει το λόγο. Λοιπόν, τώρα θα ζητήσω από τον κύριο Herbert, πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να πει ίσως δύο λόγια για το πρόγραμμα και μετά ε, να επιστρέψουμε στην κυρία Μακλάρκιν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την ε, εισηγήτρια, την κυρία Μακλάρκιν, γιατί ε, αναγνωρίζει τη σημασία του να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η ανάπτυξη μέσω των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η να γίνει μείωση της γραφειοκρατίας. Εν γέννη, συμφωνούμε με αυτά που είπαν και οι άλλοι ομιλητές. Επίσης εκτιμάμε και τις δικές σας προσπάθειες να επιτευχθούν ε, συμβιβασμοί. Η περίπτωση του τουρισμού αποτελεί καλό παράδειγμα αυτής της αίσθηση για συμβιβασμό. Περιλαμβάνει στο, ε, στη συνθήκη και πραγματικά η ανάγκη για ανάπτυξη σε κάποιες περιοχές της Ευρώπη ε, στην περίπτωση αυτές ε, ο τουρισμός είναι καλό παράδειγμα αλλά σε κάποιες τροπολογίες έχει δοθεί μια τάση που δεν ήταν η αρχικά σκοπούμενοι, δηλαδή το Enterprise Network κάνουν πολλά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά κάνουν και πολύ περισσότερο από αυτό. Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο να μην δοθεί η εντύπωση ότι το δίκτυο Enterprise Europe θα κάνει μόνο αυτό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κάνει κάτι πολύ περισσότερο από το να εντοπίζει προγράμματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα, για την εποπτεία και αξιολόγηση, βεβαίως, επί του πνεύματος συμφωνούμε, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στη διατύπωση, διότι στο κόσμο έχουμε συμπεριλάβει κάποια στοιχεία εποπτείας, επιτήρησης και πρέπει να, να αποφύγουμε στο τέλος να υπάρξουν υπερβολικά πολλά, ε, πολλές εποπτείες που θα προκαλέσουν βάρη και καθυστερήσεις. Συνολικά εκτιμούμε ιδιαίτερα την έκθεση και θέλουμε να πούμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε περαιτέρω όλα αυτά τα θέματα, εάν αυτό σας ενδιαφέρει. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κύριε Χέρβερτ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Μακλάρκιν για να ανακεφαλαιώσει και ενδεχομένως να θέσει κάποια άλλα θέματα πριν γίνει η αυριανή ψηφοφορία. Κυρία Μακλάρκιν. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα σχόλιά της. Προσπαθώ να κάνω αυτή την ε, χρηματοδότηση κόσμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμη. Να υπάρχουν λίγα βάρη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να τις βοηθήσουμε. Θέλουμε επίσης να αποτελεί κάτι το συμπληρωματικό του ορίζοντα 2020 και όχι να απομονώνονται οι επιχειρήσεις και να χρηματοδοτούνται είτε από το ένα είτε από το άλλο. Πιστεύω ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την γραφειοκρατία. Όταν μιλάω για τη, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μου περιγράφουν τεράστια βάρη γραφειοκρατικά. Θέλω να πω στην Επιτροπή, η οποία μας βοήθησε πάρα πολύ στην ευχαριστήσω εσά και τους ε, συνεργάτες σας και τους συμβούλους μου και τα μέλη της Γραμματείας ότι στο ε, Europe Enterprise ε, βεβαίως αυτό είναι ένα δίκτυο αλλά η σημασία του να επισημαίνει ε, τις δυνατότητες χρηματοδότητες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αισθάνονται ότι βρίσκονται σε ένα λαβύρινθο είναι πολύ θετικό και όσον αφορά το βάρος εποπτείας ίσως αυτό είναι για την Κομισιόν αλλά θα ήταν δύσκολο σε σχέση με την έλλειψη πρόσβασης ε, στη χρηματοδότηση. Πρέπει λοιπόν να ε, εποπτεύουμε, να παρακολουθούμε ποια είναι η κατάσταση με το δίκτυο αυτό. Για να είμαστε αποδοτικοί πρέπει να φροντίσουμε ότι ε, θα θα αποσυρθούν αυτά τα εμπόδια. Ελπίζουμε ότι θα είναι επιτυχημένη αύριο η ψηφοφορία. Ευχαριστώ όλους για την συνεισφορά σας. Ε, ευχαριστώ. πάρα πολύ για τη δουλειά που κάνατε. Ο κύριος Ρέπο σας περιέγραψε ως πολύ αποφασιστική και αυτό είναι πολύ ε, σημαντικό. Δείχνει ε, πόση, πόση προσπάθεια καταβάλλετε. καταβάλλετε. Θέλω να σας ενημερώσω ε, σχετικά με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο την ε, γνωμοδότηση του κυρίου Μπουζόη που θα πάει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Ο κύριος Μπουζόη δεν θα μπορέσει καθόλου να παρευρεθεί σήμερα το απόγευμα μόλις μάθαμε. Όμως, εξ όσων αντιλαμβάνομαι, οι σκιώδεις έχουν συμφωνήσει με τον εισηγητή για τις τροπολογίες που θα ψηφιστούν αύριο. Αυτό πρέπει να γίνει λόγω των διαπραγματεύσεων με την Επιτροπή Προϋπολογισμού και το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο θα μιλήσει με το Συμβούλιο. Ξέρω ότι είναι εδώ κάποιοι από τους Σκιώδης, ο κύριος Μπαλταζάρη, ε, ο κύριος Κόζος είναι και αυτός εδώ. Έχει κάποιος από εσά ε, κανένα σχόλιο που θα ήθελε να καταγραφεί ή σας αρκεί να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία αύριο και όλα είναι σαφή. Ο κύριος Παλτασάρη ε, μου ε, κάνει νόημα ότι όλα είναι εντάξει, εντάξει και από άλλους, ωραία. Οπότε, υποβάλλω το θέμα επισήμως και αύριο συμφωνούμε για την ψηφοφορία. Τώρα κανονικά ε, έχουμε κερδίσει λίγο χρόνο, γιατί έπρεπε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για τις ε, προτάσεις ε, για την επίλυση καταναλωτικών διαφορών και την, στις 15 ε, και 50. Μάλλον λοιπόν να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα μέχρι τις παραδέκα. Ε, ούτως ή άλλως δεν είναι εδώ οι σκιώδεις. Θα κάνουμε λοιπόν ένα πολύ μικρό ε, διάλειμμα και θα ξαναρχίσουμε αμέσως στις 4 παρα 10. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν παρα 10 με τον κύριο Κρέκ και την κυρία Τουίν για τις προτάσεις για το ΕΕΔ και το ΙΕΔ. Uh, λοιπόν, ε, είναι κανείς ε, που δεν ήταν στο πρώτο μέρος της συνεδρίασης και ήρθε τώρα για τη συζήτηση αυτών των δύο εξαιρετικά σημαντικών προτάσεων για την ε, εναλλακτική επίλυση διαφορών και την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών. Καλωσορίζω τους εισηγητές για τις δύο προτάσεις, τον κύριο Λουί Γκρέχ, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, ε, πολύ γνωστό και ως εισηγητή για την ε, εμβληματική έκθεση της ενιαίας αγοράς ε, για τους πολίτες και τους καταναλωτές που οδήγησε στην πράξη για την ενιαία αγορά. Ήταν δική μας ιδέα και ο Λούι Γκρέκ την υποστήριξε και την κυρία Ρόζα Γκρέφιν Φοντούν Χόενστάιν, η οποία ασχολείται με το θέμα των ηλεκτρονικής ε, επίλυσης διαφορών. Ο Χάνς Μάιερ είναι εδώ για την έκθεση του... Για την πρώτη έκθεση, μετά έχουμε τους σκιώθητες και για τις δύο προτάσεις, την κυρία Ρούλε και για τους δύο κύριο Φόρπες και για τις δύο προτάσεις. Και δεν βλέπω ακόμα τους υπόλοιπους σκιώδοντες. Επίσης, Χαίρομαι που καλωσορίζω από την Επιτροπή την κυρία Ζακλίν Μάινερ, Διευθύντρια Καταναλωτικών Υποθέσεων και την Κριστίνα Ρούσου, που είναι υπεύθυνη για αυτό το πολύ σημαντικό ε, θέμα. Δίνω λοιπόν, θα τους δώσω αργότερα το λόγο. Χωρίς λοιπόν περαιτέρω καθυστέρηση, καλώ τους εισηγητές να μιλήσουν ένας μετά τον άλλον και μετά θα πάμε στους σκιώδης. Θα κάνουμε συνδυαστική ε, συζήτηση και των δύο ε, εκθέσεων, οπότε ε, κύριε Κρέκ, τις τροπολογίες και τις συμβιβαστικές θα συζητήσουμε. Ελπίζω να έχετε όλοι αντίγραφα των προτινόμενων συμβιβαστικών λύσεων και τροπολογιών. Έχουν δοθεί στα αγγλικά. Τα έχετε μπροστά σας. Louis Craig. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το γεγονός ότι έπρεπε να επεξεργαστούμε πάνω από 400 ε, τροπολογίες έκανε όλη τη ε, διαδικασία αυτή ιδιαίτερα πολύπλοκη, ειδικότερα λόγω και των χρονικών περιορισμών. όλα αυτά, ε, εξαιτία τη πολύ σημαντική συνεργασία με του κυρίου Μάγερ, Όσφολτ, Ρούλε, Φόξ και Ντεόγκ, καταφέραμε να ε, συμβιβάσουμε τις ε, διάφορες ε, αποφάσεις και πέρυσι, απόψεις συγγνώμη, και την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο μπορέσαμε να καταλήξουμε σε μια σειρά σημαντικών αποφάσεων για αυτό το θέμα, ειδικότερα για το πεδίο εφαρμογής ε, σχετικά με τα, την εναλλακτική επίλυση διαφορών, την ελευθερία και την νομιμότητα, το άρθρο 6, την αμεροληψία με τον κύριο Μπουζόη, την ε, παροχή πληροφοριών στους ε, καταναλωτές, ειδικότερα θέματα για τα κράτη-μέλη, σε επαφή με τους εμπόρους και τους καταναλωτές, το κόστος της αναλεκτικής επίλυσης διαφορών και όλοι την, ε, όλο το σκεπτικό πίσω από αυτή την οδηγία που είναι μια ελάχιστη εναρμόνιση. Για να δούμε λίγο ε, σύντομα τις συμβαστικές τροπολογίες. Η 1, 2 και 4 ε, αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι αυτή θα εφαρμόζεται μόνο σε συμβατικές διαφορές εξαιρώντας ε, τις μη οικονομικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος. Δεύτερον, η ε, ε, υιοθέτηση των ελάχιστων προδιαγραφών. Παρ' αυτά, τα κράτη-μέλη μπορούν να διατηρήσουν να εγκρίνουν επιπλέον διαδικασίες σε αυτή την οδηγία. Τρίτον, το γεγονός ότι εξαρτάται από τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν αν επιβάλλεται ή προτείνεται λύση το γεγονός ότι ε, η οδηγία εφαρμόζεται βασικά για τις διαφορές μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων. Ε, το ΕΛΚ θέλει να γίνει ε, ψηφοφορία σε, τμήμα, σε τμήματα γιατί θεωρεί ότι θα ήταν αντιπαραγωγικό να πάμε και στην κατεύθυνση έμποροι προς καταναλωτές ή έμποροι προς εμπόρους και για να υπάρχει μια πραγματική αποτελεσματική εφαρμογή αυτής της οδηγίας πρέπει να παραμείνουν στην κατεύθυνση καταναλωτές προς έναντι εμπόρων. Συμβαστική τροπολογία 3 ασχολείται με τα δύο ευαίσθητα θέματα του πεδίου και της ανεξαρτησίας, όπως και με τις ε, σημαντικές διασφαλίσεις που χρειάζονται ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία ειδικότερα σε, κάποιες ειδικές, ε, σε κάποιους ειδικούς τομείς. Οι 5 και 6 έχουν να κάνουν με τον ορισμό των συμβατικών υποχρεώσεων ενώ οι 7 ε, και 8 έχουν να κάνουν με την προσβασιμότητα των καταναλωτών στην εναλλακτική επίλυση διαφορών. Από την άλλη, η συμβαστική λύση 9 αναγνωρίζει τη δυνατότητα των κρατών μελών να διατηρήσουν ή να εισαγάγουν διαδικαστικούς κανόνες ε, με την απαραίτητη δικαιολόγηση έτσι ώστε ε, μια εναλλακτική επίλυση διαφορών να απορρίψει συγκεκριμένες ε, διαφορές. Η 10 σχετίζεται με τις πληροφορίες που πρέπει να δοθούν για την εναλλακτική επίλυση διαφορών, ενώ η 11 και 12 ασχολούνται με το κόστος και το χρονικό πλαίσιο που χρειάζεται για την επίλυση των ε, διαφορών. Οι 13 και 14 ασχολούνται με τη δεσμευτική και μη δεσμευτική φύση της διαφοράς και το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών σε περίπτωση σε περίπτωση που η επίλυση είναι δεσμευτική. Οι 15 και 16 συμφιλώνουν τις διάφορες απόψεις σχετικά με τις υποχρεώσεις του εμπόρου να παράσχει πληροφορίες ε, ε, στον καταναλωτή για τους φορείς επίλυσης ε, διαφορών. Οι 16 και 17 έχει να κάνει με τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών, ενώ οι 18 ασχολείται με την με τον καθορισμό των αρμόδιων ε, αρχών για την επίλυση καταναλωτικών διαφορών. Η 19 ασχολείται με την γεωγραφική κάλυψη της ΕΕΔ, ενώ η 20 ασχολείται με το θέμα της εμπιστευτικότητας και της ιδιωτικότητας. Η τελευταία συμβαστική τροπολογία 21 αναφέρει ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με τον έμπορο όσο είναι δυνατόν πριν ξεκινήσουν ε, μια διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης διαφοράς. Η τελευταία ε, συμβιβαστική είχε να κάνει με το άρθρο 6 που είχε να κάνει με την ανεξαρτησία και μεροληψία, αλλά αποφασίσαμε με τον κύριο Μπουζόη ε, ότι σε σχέση με αυτό που είχαμε ήδη ε, αποφασίσει για το 6 που είναι αρμοδιότητα της Γιούρη και αυτό που έχει να κάνει με τις διασφαλίσεις στο άρθρο 2,8 θα συμπεριληφθούν ε, η, η τροπολογία 22 που θα έπρεπε να υπήρχε εδώ και δεν υπάρχει. Ε, κυρίες και κύριοι, ε, προσπαθούμε μέσα από τις τροπολογίες να καλύψουμε προβλήματα επαναλήψεων και ε, ασυμβατότητας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Σκιώδης, ε, το προσωπικό και την Επιτροπή για την συνεργασία τους σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Γκρέκ και για, την επισκόπηση των ε, συμβαστικών τροπολογιών. Η κυρία ε, Τιούν τώρα θα μας παρουσιάσει τις τροπολογίες για το πακέτο IDR. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους όσοι κατέθεσαν τροπολογίες. Συνεργαστήκαμε με τους Κιώδης σχετικά με αυτές τις ε, συμβαστικές τροπολογίες. Συζητήσαμε πολλές φορές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καταλήξαμε σε προτάσεις που νομίζω ότι θα ε, τύχουν της ευρύτερης υποστήριξής σας. Και αυτές τις ε, προτάσεις συμβαστικών τροπολογιών έχω ήδη δεχτεί πολλά θετικά σχόλια από τους κοιόδης, αλλά και εδώ κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Επιτροπής. Και έχω την εντύπωση ότι ε, υπάρχει ευρεία ε, συμφωνία. Το αποτέλεσμα, για να το θέσω εν συντομία, έχει ως εξής. Συμφωνήσαμε ότι η πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών που έχει ως βασικό στόχο να δώσει ένα αίσθημα ασφάλειας σε εκείνους ε, που ψωνίζουν διασυνοριακά και νιώθουν μια ανασφάλεια μέσα σε αυτή τη τζούγκλα των 27 ε, διαφορετικών κανονιστικών ε, πλαισίων των κρατών μελών, έχει ως αποτέλεσμα αυτή η πλατφόρμα, η ΕΔ, να ε, εξυπηρετεί ε, την κατεύθυνση καταναλωτές προς επιχειρήσεις αλλά και την κατεύθυνση επιχειρήσεις προς καταναλωτές όπου είναι δυνατόν σύμφωνα με την διαδικασία εναλλακτική επίλυσης καταναλωτικών διαφορών. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με θέματα ε, διασυνοριακού και εσωτερικού ηλεκτρονικού εμπορίου. Ε, θα έχει, είναι η, πλατφόρμα αυτή διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι πλήρως υπεύθυνη για τη μετάφραση. Αποφασίσαμε, και αυτό θα το δείτε τελικά στην έκθεση, ότι ε, θα είναι ε, ο κατηγορούμενος, ο εναγόμενος ο οποίος θα είναι ε, αυτός που θα αντιδρά πρώτα και ο ενάγων θα είναι ε, αυτός ε, που θα καταθέτει την πρόταση για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών. Ασχοληθήκαμε επίσης με την πλήρη ενσωμάτωσή του στο Europortal αλλά και με τη δυνατότητα πρόσβασης και μέσω άλλων οδών αν είναι δυνατόν. Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα επίλυσης, δεν την παρέχει. Επίσης, τα σημεία επαφής για την πλατφόρμα, η ΕΔΕ, θα βρίσκονται στα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών από το δίκτυο ε, Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών. Αυτά είναι τα βασικά σημεία για τα οποία νομίζω ότι θα καταφέρουμε να έχουμε ευρεία ε, υποστήριξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Τιν. Και τώρα πάμε στους σκιώδεις. Καταρχάς για το ΕΛΚ, ε, για την έκθεση ΚΡΕΚ, Hans Peter Mayer. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να πω ε, εξ αρχής ευχαριστώ και να συγχαρώ τον συνάδελφο κύριο Κρέχ όχι μόνο ε, για την εκθεσή του, είναι αυτονόητο ε, αυτό, αλλά και για το γεγονό ότι ήταν ανοιχτό σε συζήτηση και σε συμβιβασμό κατά, τη, και συμβιβασμό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σπάνια είναι να, είναι να μπορούμε να έχουμε μια καλή ε, επίλυση αυτής της διαφοράς απόψεων. Να πω ε, κάτι σύντομο, γιατί μαζί επεξεργαστήκαμε αυτές τις τροπολογίες. Ε, Είχαμε μία ε, συνεδρίαση στην οποία δεν φαινόταν αν θα τελειώναμε ή θα έπρεπε να συνεχίσουμε σε άλλη συνεδρίαση. Τελικά καταλήξαμε πολύ γρήγορα. Φαίνεται λοιπόν μια καλή συμβαστική λύση για την ψηφοφορία και με καλή πλειοψηφία για τόσο σημαντικά ζητήματα, ε, τα οποία θα ψηφιστούν. Είμαι πεπισμένος τελικά. Επίσης ανέφερε ο εισηγητής ότι έχουμε την κατεύθυνση μόνο ε, από τους καταναλωτές έναντι των εμπόρων. Αυτό δεν είναι συμβιβασμός. Εμείς ε, ε, συμφωνήσαμε ως ΕΛΚ παρόλο που δεν είχαμε αυτή την άποψη. Θα γίνει χωριστή ψηφοφορία στο σημείο 7 είπατε, όμως εμείς την αποσύρουμε γιατί δεν θέλουμε ε, εξ αρχής ε, να κάνουμε μια χωριστή ψηφοφορία για κάτι που θα δοθεί ως ε, νόμος και με αυτό θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι για συμβιβασμούς και ίσως αργότερα να συζητηθεί η ιδέα μας και να υπάρχει και θέμα επίλυσης διαφορών εναντίον από την, στην κατεύθυνση έμποροι εναντίον καταναλωτών αργότερα. Εξ αρχής λοιπόν πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μια διμερή επίλυση μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων ε, χωρίς να υπάρχει άμεσα προσφυγή στην ΕΕΔ ε, ίσως ε, πρώτα με μια πρώτη επαφή με τους εμπόρους. Αυτό επιτεύχθη ο συμβιβασμός. Από την άλλη ήταν ξεκάθαρο στόχος μας να μην ε, καταστρέψουμε τα εφιστάμενα συστήματα, αλλά να τα ενσωματώσουμε όσο γίνεται. Φυσικά, προσπαθήσαμε να διατυπώσουμε στο συμβιβασμό ότι τα συστήματα αυτά θα είναι υψηλής ποιότητας και ότι θα υπάρχει και μια κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση για αυτά. Τέλος, σχετικά με τη χρηματοδότηση, και εκεί παλέψαμε, εγώ θεωρώ ότι οι ιδιωτικές διαφορές ε, δεν θα πρέπει να πληρώνονται από τα κράτη-μέλη, αλλά να χρηματοδοτούνται και ιδιωτικά και πάλι. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη ε, υπηρεσία μέσα στα πλαίσια της ε, ε, ΕΕΔ που θα έχει να κάνει και αυτή με την επικουρικότητα ώστε αυτές οι διαδικασίες να προσφέρονται στα κράτη-μέλη είτε δωρεάν είτε με χαμηλό κόστος έτσι ώστε τα κράτη-μέλη ε, να έχουν και κατάλληλο πεδίο ώστε να μπορούν αυτό να το ρυθμίσουν νομικά. Συνολικά λοιπόν να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά Λουί Κρέκ που ήσασταν εισηγητή. Τώρα για το θέμα της ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών που ε, είναι στενά συνδεδεμένη με την ΕΔ, δεν μπορούμε να τα διαχωρίσουμε αυτά το δύο. Η κυρία Τούν μαζί μας συζήτησε, έκανε μια πολύ μεγάλη συζήτηση και προσπαθήσαμε να βρούμε μια ε, συμβαστική λύση για, για τις δύο περιπτώσεις, την εναλλεκτική επίλυση διαφορών και την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ρέπο τώρα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Τούν για την εξαιρετική συνεργασία της. Είμαι πολύ ευτυχής που βλέπω ότι θα υπάρχει σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες διαθέσιμο το έντυπο ηλεκτρονικής υποβολής παραπώνων. Εγώ εκπροσωπώ μια εξαιρετικά μικρή γλώσσα και γι' αυτό επανειλημμένος Αναφέρθηκα στο ότι ε, ανησυχώ ότι οι αυτόματες μεταφράσεις, οι μεταφράσεις που γίνονται αυτόματα έχουν ποιοτικά θέματα. Αλλά επανειλημμένως τώρα μου διαβεβαίωσαν ότι δεν θα πρέπει να ανησυχώ. Προσπαθώ να, μην ανησυχώ και ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Από την άλλη όμως πλευρά, για όλους εμάς και για τους καταναλωτές, για τους ε, κατασκευαστές, για όλους, το καλύτερο θα είναι να, να μην χρησιμοποιηθεί πολύ συχνά αυτό το σύστημα. Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο θα αναπτυχθεί και μάλιστα το διαμεθοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά επίσης ελπίζω ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα ή, εν πάση περιπτώσει, θα υπάρχουν τα λιγότερα δυνατά προβλήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο πρόεδρος, ο κ. Ρόσφορ, ο οποίος θα αναφερθεί και στις δύο προτάσεις. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε και για τις δύο ε, εκθέσεις. Ευχαριστώ και τους δύο εισηγητές που έκαναν σοβαρή δουλειά και που εισάκουσαν τις προτάσεις μας. Ε, ο κύριος Γκρέος έχει τεράστιο ταλέντο, το οποίο θα το περιέγραφα ως εξής από καιρού σε καιρό ξέρει να απομακρύνεται από την αρχική του θέση και να προχωρεί προς συμβιβασμό. Χαίρομαι, αλλά θα ήθελα και άλλοι να απομακρύνονται λίγο από την αρχική του θέση και να πηγαίνουν προς ένα συμβιβασμό. Ε, άκουσα προλίγου και τον κύριο Μάγερ που μίλησε. Θέλω επίσης να σχολιάσω το σύνολο αυτών των συμβιβαστικών τροπολογιών ε, και να αναφερθώ επιτροχάδιν σε κάποια θέματα από των οποίων θα υπάρξουν συμβιβασμοί πιο δύσκολη από ό,τι οι υπόλοιποι. Το, υπάρχει το C2B, το B2C, είναι ένα θέμα σημαντικό που το θέτουν οι διάφορες πλευρές. Ε, εγώ από πλευρά μου, όπως και ο κύριος Γκρέσ, συμφωνώ στην, εναλλακτική επίλυση διαφορών να, υπάρχει, να επικεντρωνόμαστε στο B2C. Όχι, λάθος λέει ο μιλητής, το C2B. Κάθε φορά μπερδεύομαι ο καταναλωτής είναι αυτός που έχει ανάγκη να διευθετήσει ένα θέμα. Το λέω αυτό, το λέω όχι για λόγους δογματικούς, όχι γιατί πρέπει να υπερασπιζόμαστε μόνο τους καταναλωτές και δεν θα πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχα εργαλεία για, τους, ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όχι, για την ε, το πόσο εμφανές θα γίνει αυτό. Αν θέλουμε να πούμε ότι είμαστε στην υπηρεσία της υπεράσπισης του καταναλωτή, αυτό θα είναι κάτι το πολύ ισχυρό και πολύ σωστά ε, θα εφαρμοστεί στα κράτη-μέλη. Είναι πολύ πιο ισχυρό αυτό από το να πούμε ότι ε, θεσπίζουμε ένα συμμετρικό σύστημα, γιατί για τα μάτια του καταναλωτή η συμμετρία δεν υπάρχει. Συμφωνώ λοιπόν απόλυτα με τον εισηγητή του κ. Γκρέσ ότι πράγματι αυτό που σημασία έχει εδώ είναι να διευθετηθεί τα θέματα των καταναλωτών και στο σχέδιο έκθεσης αναφέρεται ότι στα κράτη-μέλη από την άλλη πλευρά υπάρχουν και εκεί συμφέροντα, αλλά δεν θα πρέπει να τα εμποδίσουμε. Αυτό δεν είναι πιο ασήμαντο όσον αφορά την επίλυση των διαφορών, αλλά είναι πιο ασήμαντο σε σχέση με το γεγονός ότι θέλουμε να ανακοινώσουμε το σύστημα αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και χαίρομαι ε, που ο κύριος ε, Μάγερ προλίγου μας είπε ότι δεν θα ζητήσει στην τελική ε, ψηφοφορία να γίνει χωριστή ψήφος. Γιατί Υπάρχει μια, ένας άλλος συμβιβασμός στην ηλεκτρονική επίλυση γιατί η κυρία Τούν ε, επέμενε και οι δύο συνομιλητές να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το μέσο. Αυτά ήθελα να πω επ' αυτού. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γκρέσ που ως εισηγητής υπογράμμισε κάτι σημαντικό για μας, δηλαδή τους ε, διαμεσολαβητές επιχειρήσεων, όπου ενσωματώνονται σε όλους τους συμβιβασμούς, όλες τις ε, εκδοχές ε, ε, υπάρχουν αυτοί οι διαμεσολαβητές επιχειρήσεων και αυτό μας ευχαριστεί. Τώρα, στο θέμα των πληροφοριών, της ενημέρωσης, δεν αναφέρθηκα σε αυτό. Η υποχρέωση των... Ε, της είναι κάτι που συζητήθηκε το να αναφέρεται σε, σε όλα τα τιμολόγια θεωρήθηκε επιπλέον βάρος για τις επιχειρήσεις, όμως απολύτως ε, ε θεμελιώδες να είναι προσυμβατικά ε, όργανα και αυτά τα μέσα να αναφέρονται ξεκάθαρα και σαφώς. Για το γεγονός, όσον αφορά το γεγονός ότι πρέπει ο καταναλωτής όταν θέλει να χρησιμοποιήσει μια εναλλακτική διαδικασία τη διαφορών θα πρέπει να έχει εξαντλήσει την ε, χρήση της επιχείρησης πελατών, την υπηρεσία επιχείρησης εξυπηρέτησης πελατών. Συμφωνούμε με αυτό, αλλά υπάρχουν επιχειρήσεις για τους οποίες ε, ε, θα, με τις οποίες θα δυσκολευτεί ο καταναλωτής και απέναντι σε αυτή τη σχετικά δύσκολη κατάσταση θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το σύστημα που δημιουργούμε θα πρέπει από μόνο του να λειτουργήσει όταν ε, λειτουργεί μεταξύ ενός ε, δύο λογικών συνομιλητών, αλλά θα πρέπει να λειτουργεί και όταν από καιρού σε καιρό οι συνομιλητές δεν είναι απολύτως λογικοί. Θα πω δύο λόγια τώρα και για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών. Ε, πράγματι ευχαριστώ την εισηγήτρια. Θα πρέπει η πλατφόρμα αυτή να βρίσκεται και σε άλλους ιστοτόπους πέρα από το Euro Europe, να μην ε, υπάρχει πρόσβαση μόνο μέσω αυτής της πλατφόρμας. Σας ευχαριστούμε που μπορέσατε να συμπεριλάβετε την έννοια της ε, ολοκληρωμένης αντίληψης, δηλαδή όλοι οι καταναλωτές και κυρίως οι ευάλωτοι θα μπορούν να έχουν μια τέτοια προσέγγιση, θα πρέπει να μην αποκλείονται από αυτή την πλατφόρμα. Και εδώ πρέπει να υπάρχουν όλες οι αναγκαίες εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων όταν αυτές διακινούνται ηλεκτρονικά. Όπως και ο κύριος Γκρέσ, ε, θεωρώ ότι σχεδόν όλη η δουλειά έχει σχεδόν γίνει, ότι συνεργαστήκαμε μεταξύ μας πολύ καλά και ότι πρέπει απλώ να φροντίσουμε ότι αυτό το οποίο αποτελεί μια πρόοδο για τις αγορές, για την εσωτερική αγορά και για τους καταναλωτές ε, θα καταφέρει θα καταφέρουν τα κράτη-μέλη και η Επιτροπή να το κάνουν απολύτως συγκεκριμένο για να είναι εφαρμόσιμο και χρήσιμο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Μετά από την θετική σας προσέγγιση και υποστήριξη κυρία Ρουίλε. Δεν θα πω κι εγώ πολλά. Ευχαριστώ και τους ε, δύο εισηγητές. Ήταν πολύ καλή η συνεργασία. Το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό. Υποστηρίζω πλήρως τους συμβαστικές τροπολογίες εξ αρχής ε, ε, για την ε, τελευταία τροπολογία για το άρθρο 5 είχα κάποιες επιφυλάξεις αλλά έχουμε μια διατύπωση τέτοια που να μην οδηγεί σε δίκη αλλά να ασκεί πίεση ώστε να προσπαθεί κανείς εκ των προτέρων να επιλύσει το πρόβλημα. Επίσης, για το θέμα των εμπόρων καταναλωτών συνήθως ε, ε, αυτές οι διαφορές ε, που προκύπτουν έχουν να κάνουν με καθυστερήσεις πληρωμών ή μη παράδοση προϊόντων. Και αυτό σημαίνει σημαντικό πρόβλημα και γι' αυτό θα ήταν και γι' αυτό είναι καλό για μας που σε αυτή την περίπτωση, σε αυτό το πρώτο στάδιο περιοριζόμαστε στην κατεύθυνση C2B. Επίσης υπάρχουν συστήματα στους τομείς αυτούς που διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Ε, σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει αποζημίωση. Το βρετανικό σύστημα, για παράδειγμα, είναι τελείως διαφορετικό από ό,τι σε άλλα κράτη-μέλη. Ε, και ε, βρήκαμε λοιπόν μια λύση η οποία ε, δεν ε, θα θέτει υποαμφισβήτηση τα υφιστάμενα συστήματα αλλά ασκεί πίεση στα κράτη-μέλη να γίνουν πιο ενεργά σε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστώ πολύ τους εισηγητές και συντάσσομαι πλήρως μαζί τους για την επίλυση που, για, τις συμβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Και τέλος ο κύριος Φόξ από τους Σκιώδης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να αρχίσω με την εναλλακτική επίλυση και να ευχαριστήσω τον κύριο Γκρέχ και όλους τους εμπλεκόμενους. Παρά τις ε, στενές προθεσμίες φτάσαμε σε συμβιβασμούς που θα οδηγήσουν σε προστιθέμενη αξία στην αγορά. Η ομάδα μου συμφωνεί με τις τροπολογίες συμβιβασμού, αλλά σε τρεις τομείς ε, θα ήθελα να εκφράσουμε ανησυχίες. Στο Σύμβασμο 9 θα ήθελα ο εισηγητής ε, να αποσύρει την προαπέτηση των 14 ημερών. Και νομίζω ότι η απάντηση, θα πρέπει να δοθεί απάντηση στον καταναλωτή εν ευθέτω χρόνο. Αλλά οι 14 μέρες δεν θα μπορέσουν να ισχύσουν έμπρακτα και άρα θα πρέπει να πούμε, μάλλον γράψουμε promptly, εν χρόνο, έτσι ώστε να υπάρχει μια αναλογικότητα. Στον Σύμβασμο 14 θα ήθελα μια μικρή αλλαγή του 9β, δηλαδή με βάση τις απαιτήσει του καταναλωτή. Αυτό να αναφέρουμε, διότι ανταποκρίνεται στην αιτιολογική σκέψη 21C. Και άρα το 9B θα αναφέρει ότι τα κράτη-μέλη θα διασφαλίσουν έτσι ώστε να βρεθεί μία λύση από πλευράς καταναλωτή. Και στη συνέχεια και η συνέχεια του άρθρου παραμένει η ίδια. Τέλος. 15 και 16 συμβιβασμοί. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι και νομίζω ότι πρέπει να θέσουμε όρους στους εμπόρους για να δούμε τι καλύπτεται στα πλαίσια του ADR, της εναλλακτικής επίλυσης διαφόρων. Πολλές φορές όμως υπάρχει, επιβάλλεται φόρτο στους εμπόρους και οι καταναλωτές έχουν έχουν την εντύπωση ότι ο έμπορος θα χρησιμοποιήσει αυτούς τους φορείς. Θα ήθελα οι κύριοι Γκρέχ και άλλοι σκιώδεις να το δουν αυτό το θέμα. Ως προς την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κυρία Τουν για την εργασία που επιτέλεσε. Οι εισηγητές δέχτηκαν πολλά στοιχεία και υποδείξεις μας και η ομάδα μας, η ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών μπορεί να δεχτεί την πρόταση της ηλεκτρονικής επίλυσης. Ευχαριστούμε κύριε Φόξ. Υπάρχουν άλλοι βουλευτές που θα ήθελαν κάτι να προσθέσουν. Ο κύριος Σφάμπ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Από τη δική μου πλευρά και ως προς τη γενική αυτή συζήτηση θα ήθελα και εγώ να υποστηρίξω την ιδέα ότι μπορούμε να περάσουμε αυτές τις δύο προτάσεις πριν από την καλοκαιρινή διακοπή. Γιατί και για την ενιαία αγορά και για την Επιτροπή είναι πολύ σημαντικό για μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Hans Peter Mayer για τις προσπάθειες που κατέβαλε. Μιλήσαμε και για το γλωσσικό καθεστώ σήμερα με την κυρία Τιν όταν μιλήσαμε για το σύστημα πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς. Οι δυνατότητες μετάφρασης είναι πολλές φορές περιορισμένες και οι υπηρεσίες δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν μέχρι τούδε. Αλλά και στην περίπτωση το, της ηλεκτρονικής επίλυσης υφίσταται αυτό το ζήτημα. Όπως είπε η κυρία Τιν, χρειαζόμαστε ένα μακρόπνο, μακροχρόνιο σύστημα το οποίο να είναι λειτουργικό. Και ελπίζω αυτό να απασχολεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να μην το αφήσουμε δηλαδή, να το βάλουμε στην άκρη. Εάν δεν υπάρχουν άλλοι ομιλητές, θα ήθελα η κυρία Μάινερ να σχολιάσει, η κυρία, η κυρία Ρουσό, η κυρία Μάινερ, δεν ξέρω ποια θα μιλήσει πρώτα. Η κυρία Μάινερ θα αρχίσει και θα θέλαμε να, να ακούσουμε τα σχόλιά σας και μετά οι Τιν και Γκρέχ θα απαντήσουν. Κυρία Μάινερ, ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους Γκρέχ και Τιν, τους δύο εισηγητές, για την εξαιρετική τους εργασία. Με μεγάλη χαρά συνεργαστήκαμε από κοντά και ε, παράλληλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Κιώδης καθώς και όλα τα μέλη αναγνωρίζουμε ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος, ιδιαίτερα αυτή τη χρονική στιγμή. Και σας ευχαριστούμε επειδή ε, συμβιβαστήκατε, επειδή δεσμευτήκατε ως προς ένα χρονοδιάγραμμα, το οποίο και τηρήσατε. Η Επιτροπή αντιμετωπίζει θετικά και τις δύο εκθέσεις, καθώς και την ενδεχόμενη έκβαση των συμβιβαστικών προτάσεων. Βεβαίως θα πρέπει να εξετάσουμε τα κείμενα ενδελεχώς και να δούμε και τις δύο προτάσεις της εναλλακτικής επίλυσης και της ηλεκτρονικής εναλλακτικής. Θεωρούμε το πακέτο είναι πολύ καλό. Χαίρομαι διότι ε, κρατήσαμε τις αρχικές δεσμεύσεις. Έγινε συζήτηση για τις καταγγελίες εμπόρων κατά καταναλωτών και θα ήθελα να πω ότι στο βαθμό του δυνατού και εάν το προβλέπουν τα εθνικά συστήματα, οι καταγγελίες αυτές μπορούν να παραμείνουν και τα κράτη-μέλη μεταφέροντας την οδηγία περί εναλλακτικής επίλυσης μπορούν να επεκτείνουν τις καταγγελίες των επιχειρήσεων κατά των καταναλωτών. Στη συνέχεια θα πρέπει να αναθεωρήσουμε την οδηγία για να δούμε κατά πόσο μπορεί να επεκταθεί, αλλά δεχόμαστε τους, ε, τους λόγους, το αιτιολογικό, το αιτιολογικό του κυρίου Ροσφόρ ιδιαίτερα, σε σχέση με την περιορισμένη εμβέλεια των ε, καταγγελιών που προέρχονται από τους καταναλωτές. Ε, απογοητευτήκαμε ως προς τις ε, προαπαιτήσεις πληροφοριών γιατί απομακρυνθήκατε από την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα πρέπει να δούμε τις διασφαλίσεις που εισαγάγονται για, την, για τους ανεξάρτητους, την ανεξαρτησία των φορέων εναλλακτικής επίλυσης και θα θέλαμε να δούμε και διαδικαστικούς κανόνες που ανέφερε ο κύριος Φόξ. Θα θέλαμε να υπάρχει η βέλτιστη δυνατή λειτουργία ως προς την ηλεκτρονική επίλυση διαφόρων. Υποστηρίζουμε τις τροπολογίες ε, για την χρήση της πλατφόρμας, η οποία να είναι φιλική, ευφύης και διαφανής για τους καταναλωτές, καθώς και ασφαλής. Ως προς το γλωσσικό, καταλαβαίνω την ανησυχία του κυρίου Σφάμπ και εμείς Έχουμε προβάλει αυτό το θέμα σε μία τεχνική ομάδα για θέματα μετάφρασης και πιστεύω ότι πριν ισχύσει η πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών θα έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο υπηρεσιών στο ύψος των προσδοκιών των καταναλωτών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Επιτροπής και ιδιαίτερα τους συζητητές Γκρέφ και Τιν Εκτιμούμε την εργασία αυτή καθώς και την ποιότητα της εργασίας σας. Ωραία. Ο κύριος Γκρέχ ε, θα ήθελε ίσως να σχολιάσει καταρχήν και μετά θα δώσω το λόγο στην κυρία Τιν. Εντάχει, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Σκιώδης. Νομίζω ότι ήταν πρόθυμοι να φτάσουμε σε συμβασμούς, γι' αυτό ε, και στο τέλος το καταφέραμε. Ως προς τη σύσταση του κυρίου Φόξ, ο συμβασμός 14 μπορεί να με βρει σύμφωνο. Ως προς την 9 θα πρέπει να τη συζητήσω με άλλους ε, σκιώδεις, γιατί πρόκειται για μια ειδική σύσταση από άλλο σκιώδη και θα ήθελα τη δική του συμφωνία. Κατανοώ αυτά που λέτε, αλλά θα πρέπει να συμφωνήσει και ο άλλος σκιώδης. Ως προς το, τα 15 και 16, τις δύο προτάσεις συμβασμού θα είναι πιο δύσκολο να γίνουν αποδεκτές. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αυτά είναι και τα τελικά μου σχόλια. Η κυρία Τούν και εγώ να σας ευχαριστήσω όλους για τα ενθαρρυντικά σας σχόλια και θα ήθελα να πω ότι όταν μου ανατέθηκε αυτή η έκθεση δεν μπορούσα να φανταστώ τόσο παθιασμένες και ζωηρές συζητήσεις και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και με πολλούς εμπλεκόμενους φορείς. Αυτό ήταν άκρος ενδιαφέρον και έμαθα πολλά από αυτή τη διαδικασία αποτέλεσμα μετά από αυτό το input μας οδηγεί σε ένα εκτενές, σαφές κείμενο με επιμερισμό ευθυνών και ελπίζω και οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις να, θεωρεί, να θεωρήσουν αυτούς ασφαλείς, ιδιαίτερα ως προς τις επιγραμμικές συναλλαγές ενδοευρωπαϊκά. Δεν θέλουμε να αποκλείσουμε και την εναλλακτική την ADR, τη διαδικασία ADR. Ένα μόνο σε ένα μόνο θέμα θα ήθελα να σταθώ. Πολλοί συνέταξαν ε, τροπολογίες για την ηλεκτρονική επίλυση και όχι για το ADR. Και επειδή θα πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός, ε, τις ε, ξεχώρισα ξεκινώντας με τη 19 ε, τη δική μου. Δηλαδή θέματα ADR θα πρέπει να αφορούν μόνο την εναλλακτική επίλυση και όχι την επιγραμμική. Ε, να δούμε τις προθεσμίες και όλα τα συναφή ξεχωριστά. Έτσι ώστε να μην υπάρχουν ε, διαφορετικές απαιτήσει. Και πρότεινα έβαλα ένα πλήν στον κατάλογο ψηφοφοριών εκεί που δεν μπορώ να αποδεχτώ τις τροπολογίες. Αυτό ε, το λέω προς τους σοσιαλιστές, γιατί νομίζω ότι την χάνω ευρείας ε, υποστήριξης. Θα φτάσουμε σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ήμουν απόλυτα σαφής, το ελπίζω. Ε, θα ήθελα και πάλι να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς όλους. Και με συγχωρείτε γιατί ήμουνα ε, πολύ δύσκολη διαπραγματεύτρια, ιδιαίτερα στην κοινή μας εργασία. Και αυτό το λέω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, πρέπει να είναι κανείς και επικριτικός και επικοδομητικός. Καλή η έκβαση λοιπόν και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πάντες, λέει ο πρόεδρος, διότι πολλά επιτελέστηκαν και βλέπουμε πώς γίνεται η προπαρασκευαστική διεργασία και αποτίμηση για να δούμε πώς διαμορφώνεται και η τελική πρόταση. Αύριο λοιπόν θα ψηφίσουμε και επί των δύο προτάσεων. Δεν ξέρω κατά πόσο ο κύριος Γκρέχ και ε, άλλοι θα ήθελαν να δεχτούν τις τροπολογίες Fox και άλλων. Εν πάση περιπτώσει το αποτέλεσμα θα είναι θετικό και η Κυπριακή Προεδρία θα μας μιλήσει για αυτή την πρόταση. Αλλά αυτό θα το αφήσουμε στους δύο εισηγητές ως προς την άποψή τους για το πώς θα προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας. Άρα τελειώνουμε με τα θέματα της εναλλακτική ε, επίλυσης και της επιγραμμικής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τις κυρίες Μάιερ και Ρουσό. Ωραία. Λοιπόν, επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί από το ADR, από την εναλλακτική επίλυση. Θα ήταν σκόπιμο να αποχωρήσετε όσοι θέλετε και να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα με εισηγήτρια την κυρία Πιέτη Κάινεν. Λοιπόν, παρακαλώ, παρακαλώ αποχωρήστε όσοι είναι να αποχωρήσετε σύντομα.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 Uh, Ωραία. Σας παρακαλώ ας συνεχίσουμε, λέει ο Πρόεδρος, στο επόμενο θέμα που είναι η γνωμοδότηση για τα δικαιώματα των επιβατών σε όλους τους τρόπους μεταφορά. Η κυρία Πέτη Κάινεν είναι η συγγήτρια επί του θέματος. Έχουμε και τους σκιώδεις παρόντες. Θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Άννα Χέντ η, την κυρία Παρβάνοβα δεν τη βλέπω, ούτε του Στουν και Μπίλαν. Άρα Χέντ και Κάινεν θα κάνουν ολόκληρη, θα επιτελέσουν την εργασία αυτή, θα μας βοηθήσουν στο έργο μας. Δίνω το λόγο στην κυρία Κάινεν για να μας παρουσιάσει τις τροπολογίες πριν ε, ψηφίσουμε. Κυρία Κάινεν. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη διότι το κείμενο συμβιβασμού έφτασε πολύ αργά και η έκδοση που έχετε μπροστά σας, ο πίνακας που έχετε μπροστά σας, δεν είναι και ο τελευταίος. Θα πρέπει να λάβετε τον τελευταίο μέσα στο επόμενο λεπτό. Οι σκιώδεις έχουν τους τελευταίους συμβιβασμούς ε, μερικοί είναι τεχνικής υφής και άλλοι κινούνται επί της ουσίας. Ε, ζητώ συγγνώμη γιατί πολύ αργά σας έδωσα αυτά τα στοιχεία. Σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ καλή συνεργασία με τους Σκιώδης και με άλλα μέλη της Επιτροπής. Νομίζω ότι μας βοήθησαν ιδιαίτερα τα σχόλια και οι τροπολογίες σας για τη σύνταξη αυτών των προτάσεων συμβιβασμού, γιατί προσπάθησα να υποβάλω τα περισσότερα δυνατά στοιχεία. Αρχίζουμε με τον πρώτο συμβιβασμό που προέρχεται από εσάς και σχετίζεται με τη σημασία των καταναλωτών, δηλαδή να την χάνουν ίσης προστασίας Ξέρω ότι αναφέρεστε σε ελάχιστες προδιαγραφές, δηλαδή το ελάχιστο επίπεδο που θα μπορέσουμε να προωθήσουμε. Θεώρησα λοιπόν ότι οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα ελάχιστης προστασίας. Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά έναν ολοκληρωμένο κανονισμό ή διευθέτηση των δικαιωμάτων των επιβατών. Κατάλαβα ότι δεν υπάρχει πολιτική συνένεση και γι' αυτό χρειάζεται περισσότερη ολοκλήρωση για τα δικαιώματα των επιβατών ως προς τα διάφορα μέσα μεταφοράς και αναφερόμαστε στο γεγονός ότι θα πρέπει να έχουμε μία ολοκληρωμένη προσέγγιση των δικαιωμάτων των επιβατών. Επίσης αναφερόμαστε και στα επόμενα βήματα που θεωρούν ότι θα πρέπει να γίνει περισσότερη έρευνα έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα και μοναδικό κανονισμό για τα δικαιώματα των επιβατών. Και το could το άλλαξα στο should be carried. Θα πρέπει δηλαδή να διενεργηθεί αυτή η μελέτη και θα δούμε ποια θα είναι και η έκβαση του όλου εγχειρήματο. Ένα άλλο σημείο όπου είχαμε λεπτομεριακές ε, τροπολογίες αφορά την διαφάνεια επί των τιμών και εδώ έχουμε λάβει υπόψη και τις δικές σας προτάσεις. Και τέλος είχαμε νέες διατυπώσεις σε σχέση με κυρώσεις και αντισταθμίσεις καθώς και αποζημιώσεις που έχουν συμπεριληφθεί. Το δεύτερο σημείο όπου υπάρχει διχογνωμία έγκυται στο κατά πόσον πρέπει να ενισχύσουμε το ρόλο των ε, κέντρων καταναλωτών έτσι ώστε να έχουν περισσότερους πόρους και ε, ολοένα και αυξανόμενο ρόλο στην επίλυση διαφορών μέσα στα πλαίσια των μηχανισμών επίλυσης και κατά πόσο θα έπρεπε να έχουμε έναν πανευρωπαϊκό φορέα βοηθείας, εν είδη helpline, σε όλες τις επίσημες γλώσσες των ευρωπαϊκών κοινοτήτων, δηλαδή www.travel.eu σε μία και μοναδική διεύθυνση ιστότοπο. Υπάρχει μία άλλη γνώμη που δεν περιλαμβάνεται εδώ και που αναφέρει ότι αυτό το ζήτημα θα πρέπει να επιληθεί με καλύτερη συνεργασία των εθνικών αρχών και εθνικών ιστοτόπων. Τέλος, Πρόεδρε, είχαμε μία σειρά τροπολογιών Ε, που αφορούν τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Εδώ προσπαθώ να εντάξω αυτή την κατηγορία σε ένα συνεκτικό πακέτο έτσι ώστε να έχουμε την κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση αυτών των ατόμων, να υπάρχει σωστή αρρωγή πολιτικές ασφαλείας και να, υπάρχουν, να υπάρχει εναρμόνιση επιθεμάτων κινητικότητας και ιατρικών θεμάτων. Τα, τα δεδομένα θα πρέπει να είναι προσβάσιμα σε όλους και οι επιβάτες στη συνέχεια δεν θα πρέπει να επομισθούν επιπρόσθετα έξοδα αν εντάσσονται σε αυτές, σε αυτές τις κατηγορίες των ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα. Ούτε θα πρέπει να επομίζονται επιπρόσθετα ιατρικά έξοδα. Αυτά ακριβώς καλύπτονται και πιστεύω δεν θα υπάρξουν μεγάλες πολιτικές διαμάχες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ολοκληρωμένη αυτή παρουσίαση. Πολλέ καινούργιες ιδέες συμπεριλαμβάνονται εδώ που ελπίζω να τις λάβει υπόψη η Επιτροπή Μεταφορών. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Χέντ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Πίτα Κάνεν για την εξαιρετική συνεργασία της. Συνεργαστήκαμε πολύ καλά μαζί για αυτό το θέμα. Δεν έχω πάρα πολλά να προσθέσω τα δικαιώματα των επιβατών είναι προφανώς πολύ σημαντικά. Για μία ακόμα φορά πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι εδώ το θέμα αφορά κυρίως τους καταναλωτές. Είναι σημαντικό να αισθάνονται ασφαλείς οι καταναλωτές όταν ταξιδεύουν και ελπίζω ότι στο μέλλον θα έχουμε περισσότερο λόγο στην ομοθεσία αυτή των δικαιωμάτων των επιβατών. Όσον αφορά τις τροπολογίες, Είμαι ιδιαίτερος ικανοποιημένη επειδή μπορέσαμε να, συντάξουμε την συμβαστική τροπολογία 1, η οποία προσφέρει υψηλό επίπεδο προστασίας στους καταναλωτές. Τίποτα άλλο δεν έχω να προσθέσω παρά μόνο να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ, η κυρία Πατπάνομα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και εγώ χαίρομαι που μπορώ να πω ότι οι τροπολογίες ε, για την, ε, έχουν ε, σκοπό την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών, οι οποίες καλύπτουν πολλούς τομείς, μεταξύ των οποίων τα ένδικα δικαιώματα αυτών οι οποίοι θέλουν, έχουν προβλήματα κινητικότητας, Υπάρχουν και οι προτάσεις που στοχεύουν στην ε, εξασφάλιση της ε, ε, χρήσης όλων των μεθόδων μεταφορών όμως η γνωμοδότηση δεν νομίζω ότι είναι ο κατάλληλο σημείο να ασχοληθούμε με αυτά τα θέματα. Πιστεύω ότι τα δικαιώματα των τουριστών θα πρέπει να αντοπιστούν ως, ως ακέραιο μέρος των δικαιωμάτων των επιβατών και να μην υπάρξουν ιδιαίτερες ε, διατάξεις για αυτούς. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Πετικάνεν για το σχέδιο συμβαστικών τροπολογιών, οι οποίες καλύπτουν τα βασικά θέματα που όλοι μας θέλουμε να τομίσουμε και οι συμβαστικές τροπολογίες ε, έχουν κάνει το κείμενο πιο δομημένο και λιγότερο, ε, έχουν λιγότερες επαναλήψεις. Επίσης επαναλαμβάνω ότι τα δικαιώματα των επιβατών είναι σημαντικό κομμάτι των δικαιωμάτων των καταναλωτών και γι' αυτό πιστεύω ότι έχει πολύ σημαντικό σημαντικό ρόλο η Επιτροπή σε περαιτέρω αναθεώρηση του κανονισμού 261. Θα πρέπει ο ρόλος αυτός να αναγνωριστεί και ελπίζω αν δεν είμαστε η καθήλυνα αρμόδια Επιτροπή τουλάχιστον να είμαστε ε, ε, ε επίσης ε, όρις με την Επιτροπή Μεταφορών στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Παρβάνοβα. Οι διερμηνείς μου έκαναν νόημα ότι θα θέλανε να μιλάτε λίγο πιο αργά. Δεν σας διέκοψα όμως, ε, σας το λέω εκ των υστέρων. Η κυρία, η κυρία Τούν, η οποία είναι σκιώδης για την ομάδα των Πρασίνων. Δεν έχω να προσθέσω πάρα πολλά. Δύο λόγια. Ήταν καλή αυτή η συνεργασία μας. Καλός ο συμβιβασμός, έλεγξα μόλις την τελική του εκδοχή, τα περισσότερα σημεία καλύπτονται. Είχαμε την ιδέα του ενιαίου εισιτηρίου, που ακόμα δεν υπάρχει, το οποίο θα πρέπει να θεωρηθεί ως όραμα της Ευρώπης. Κάποια στιγμή να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε ένα πραγματικά ε, ολοκληρωμένο χώρο, χώρο επιβατών. Μας ικανοποιούν όμως οι συμβιβαστικές προτάσεις. Στην τελική έκθεση θα τις συμπεριλάβουμε και πιστεύω ότι δώσαμε έμφαση σε κάποια θετικά στοιχεία, όπως τα θέματα των επιβατών με μειωμένη κινητικότητα και τα θέματα της ενημέρωσης και το θέμα της διαφάνειας των τιμών. Χάρηκα γι' αυτό γιατί εξακολουθεί να είναι σοβαρό πρόβλημα. Συνολικά είμαστε υπέρ και θα το κάνουμε αυτό, με τα, θα ψηφίσουμε υπέρ με τα χαράς. Ελπίζουμε ότι θα περάσει και από την Επιτροπή Μεταφορών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άλλο μέλος, κάποιος άλλος που θα ήθελε το λόγο. Οπότε, ο κύριος Κόλσον νομίζω εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάρτε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο λόγια μόνο. Σημαντικό για μας ήταν οι, τα, τρόποι μεταφοράς, τα δικαιώματα των επιβατών στις διάφορες, στους διάφορους τρόπους μεταφορών να έχουν τη μορφή μιας προοδευτικής σύγκλησης και αυτό φάνηκε από τις τροπολογίες, τις συμβαστικές τροπολογίες. Πέραν αυτού, συμφωνούμε με τις περισσότερες προτάσεις που ακούστηκαν. Όσον αφορά τις τροπολογίες για τους τουρίστες, θεωρούμε ότι δεν είναι αυτό το σημείο, ε, αυτή η έκθεση στην οποία θα πρέπει να εμφανιστούν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Okay. Πρόεδρος, πολύ καλά λοιπόν. Προς το παρόν όμως θα τις ε, λάβετε υπόψη Έγινε μια συζήτηση προηγουμένως για τον τουρισμό σήμερα. Η κυρία Πιετικάνεν, θέλετε να απαντήσετε σε κάποια από τα σχόλια που ακούσατε. Σας ευχαριστώ όλους για τα θετικά σας σχόλια. Μόνο στο θέμα των τροπολογιών που δεν καλύπτουν, ε, δεν καλύπτει ο συμβιβασμός, θα αναφερθώ στο μονοψήφιο που δεν καλύπτεται από το συμβιβασμό. Τα βασικά πολιτικά πλήν είναι στην 47 και στην 38. Κανένα από αυτά τα θέματα δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ε, στο πλαίσιο των δικαιωμάτων των επιβατών, κατά τη γνώμη μου. Πρέπει να υπάρξει χωριστή νομοθεσία για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους όσοι ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό. Θα, η ψηφοφορία θα γίνει αύριο το πρωί. Πολύ ωραία. Οπότε, ο χρόνος είναι ακριβώς ο σωστός. Περνάμε στο επόμενο θέμα για την σκοπιμότητα της εισαγωγής ομολόγων σταθερότητας. Ο προφέσορ de Campos είναι ο εισηγητής, ο Βεχέν, είναι σκιώδης, ο κύριος Σμιτ δεν είναι εδώ, η κυρία Τούρνεν είναι εδώ, ο κύριος Φόξ δεν είναι εδώ, αλλά μπορεί να επανέλθει. Ο κύριος Γούσταυσον δεν είναι εδώ. Εν πάση περιπτώσει, η απαρτία των ε, σκιωδών είναι καλό, καλή. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο στον κύριο Κορέιρα Ντεκάμπο, τον καθηγητή Κορέιρα Ντεκάμπο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόκειται για μία γνωμοδότηση εδώ για τη σύνταξη κανονισμού με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη βιωσιμότητα, τη σκοπιμότητα εισαγωγής ε, ομολόγων σταθερότητας. Και από ό,τι φαίνεται, θα ήταν ε, εύκολο να φτάσουμε, φαινόταν ότι θα ήταν εύκολο να φτάσουμε σε συνένεση, αν και δεν ήταν καθόλου εύκολο τελικά. Βεβαίως δεν είναι και αδύνατον. Εργαστήκαμε με όλες τις ομάδες την ε, προηγούμενη εβδομάδα και φτάσαμε σε, στην 1, 2 και 3 πρόκειται για προτάσεις συμβιβασμού και αυτό αφορά αρκετές ομάδες. Αυτές οι τροπολογίες συμβιβασμού έχουν οριστεί και έπρεπε να εγκρίνουμε δύο προφορικές που ε, υποβλήθηκαν από την κυρία Φερχάιεν και από τον Όλε Σμιτ. Υπήρξαν ορισμένες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις δύο αυτές προφορικές, αλλά εργαστήκαμε επί αυτών των δύο και μπορούμε να πούμε έμπρακτα ότι Οι διαφορές μας ε, δεν είναι πια δυσεπίλητες. Νομίζω θα μπορέσουν να εγκριθούν οι τροπολογίες συμβιβασμού. Δεν ξέρω κατά πόσο όλοι οι σκιώδεις είναι παρόντες, αλλά θα ήταν σκόπιμο να ξέρουμε ποια είναι η θέση μας σε σχέση με τις άλλες τροπολογίες δεν ξέρω κατά πόσο είναι σκόπιμο να μπω σε λεπτομέρειες. Έχω την εντύπωση ότι δεν χρειάζεται. Δεν ξέρω κατά πόσο θα το θέλατε. Τώρα, αυτή τη στιγμή διανεμήθηκε το κείμενο, ένα κείμενο, κοινή πρότασης ε, σοσιαλιστών και ΕΛΚ σε σχέση με τις ε, προφορικές, με τις δύο προφορικές. θέματα τα οποία επιλήθηκαν τώρα εδώ την τελευταία στιγμή. Εδώ θα παραμείνω. Οι σκιώδεις μπορούν να εκφραστούν και να μου πούνε τι άποψη έχουν. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί είχαμε μεγάλες ε, ανταλλαγές απόψεων. Όλοι υποχωρήσαμε και εμείς υποχωρήσαμε σε μία από τις βασικές προτάσεις συμβιβασμού γιατί θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να προωθήσουμε ένα μήνυμα το οποίο να μην είναι αμφίγνωμο. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω του Σκιώδης και το προσωπικό που μας βοήθησε και δεν νομίζω ότι έχω να προσθέσω κάτι άλλο σε αυτή τη φάση των εργασιών, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Φερχάιεν. Να δώσω δίκιο στον προλαλήσαντα για κάποια θέματα. Είπε ότι ήταν ε, δύσκολες οι διαπραγματεύσεις και υπήρχαν ε, διχογνωμίες σχετικά με τις προϋποθέσεις πλαίσιο και τις επιπτώσεις ε, των ευρωομολόγων. Υπήρχε γενικά μια πολιτική συζήτηση και διχογνωμία και τελικά καταλήξαμε σε μια δύση, η οποία, λύση που έγινε αποδεκτή από όλους. Σχετικά με τις προφορικές ε, τροπολογίες ε, από τον Όλε Σμιτ ε, δεν υπάρχει ε, κάποια συγκεκριμένη ε, επιταγή για το τι πρέπει να γίνει. Επίσης, να πω ότι υπάρχουν πολλές ε, απόψεις σχετικά με τις επιπτώσεις και τους όρους ε, αυτών των ομολόγων. Αυτό που πρέπει να φανεί ξεκάθαρα από το κείμενο είναι ότι ε, ε, πρέπει να υπάρχουν κριτήρια που πρέπει να πληρούνται και αυτό εξ αρχής το έθεσα με τις τροπολογίες να μην γίνει κάτι προώρο χωρίς ε, να τεθούν κριτήρια. Να υπάρχει δηλαδή μια θετική διατύπωση, αλλά να, υπάρχουν, να αναφέρεται και το γεγονός ότι χρειάζονται όροι για αυτά τα ομόλογα σταθερότητας, έτσι ώστε να είναι οι επιπτώσεις τους ε, σωστές. Επίσης, οι διαπραγματεύσεις συχνά οδηγούν στο να αφήσει κάτι ε, κάποιος από τις θέσεις του. Πολλές φορές να γίνεται αυτό ε, για να μπορέσουμε να έχουμε συμβιβασμό ε, και θεωρώ ότι ε, συνολικά καταφέραμε να βρούμε μία λύση που κάπως συμβιβάζει όλες αυτές τις διάφορες θέσεις και στα κράτη-μέλη γιατί υπάρχουν διάφορες απόψεις ε, και διαφορετικές θεωρήσεις στη συζήτηση σχετικά με την εισαγωγή των ομολόγων σταθερότητας και στους πολίτες και πρέπει να προσπαθήσουμε σε όλα τα επίπεδα να υπάρχει η κατάλληλη προετοιμασία έτσι ώστε ε, ο δρόμος που θα περιγράψουμε να εξασφαλίσει μόνιμη εμπιστοσύνη στους μηχανισμούς ε, και να μην αντιδράσουν με ένταση οι αγορές ε, όταν υπάρχουν αυτά τα ομόλογα αλλά δεν υπάρχουν μηχανισμοί ε, που και έχουν γίνει με λάθος ε, deals. Θα πρέπει λοιπόν γενικώ να μπορέσουμε να θέσουμε τέτοια κριτήρια ώστε να επαναφέρουμε την εμπιστοσύνη των αγορών και να αυξήσουμε την οικονομική αποδοτικότητα, γιατί δεν είναι τα ευρωομόλογα που θα αντιμετωπίσουν την κρίση. Ε, είναι οι όροι που συνδέονται με αυτά, αλλά αποτελούν γενικά όλα αυτά ένα μέσο το οποίο θα οδηγήσει στη σταθεροποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν είναι σίγουρα το μέσο το οποίο από μόνο του μπορεί να δράσει, πρέπει να υπάρχει συνδυασμός με όρους, αλλά και με μια πιο εμβαθυμένη πολιτική, με κριτήρια και μια καλύτερη διάρθρωση των οικονομικών υπηρεσιών και της οικονομικής δύναμης, έτσι ώστε κάθε κράτος μέλος να αναλαμβάνει ε, τις ευθύνε του. Φυσικά θα υπάρχει αλληλεγγύη, αλλά πρέπει να υπάρχουν και τα κριτήρια. Ευχαριστώ πολύ τους Σκιώδης για την ε, εντατική και πολύ καλή συζήτηση και τον συγγητή που κατάφερε να ε, συνδυάσει όλες αυτές τις απόψεις και να μπορέσουμε σε πολλά σημεία να βρούμε καλές συμβαστικές λύσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, Θα αφήσω τον κύριο Σμιτ να ενημερωθεί και θα δώσω το λόγο στον κύριο Τούρνον ε, πρώτα. Ε, κύριε Τούρνον, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είμαστε ακριβώς ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, πιστεύω. Το αποτέλεσμα αυτό είναι πιο αδύναμο από αυτό της Επιτροπής Οίκων ή από τη θέση που ήδη εγκρίθηκε ε, η θέση του ΕΛΚ που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του ΤΟΥΠΑΚ. Για μένα δεν προσθέτει τίποτα. Ε, Ιδίω αν είναι κανεί υπέρ του, των ομολόγων σταθερότητα, των ευρωομολόγων ή το όπω Έτσι, λοιπόν, υπάρχει τώρα ένα θέμα των ε, ε, τα αδύναμα κράτη και αδύναμα τράπεζες. Πάμε πολύ κοντά στην άκρη του γκρεμού μετά το τελευταίο ε, διάσκεψη κορυφή και πάλι τα επιτόκια έχουν ανεβεί σε επίπεδα άνω αυτών που ήταν πριν και δεν πρέπει να στείλουμε ισχυρά πολιτικά ε, μηνύματα τα οποία αυτό το οποίο στέλνουμε με αυτό δεν είναι ισχυρό πολιτικό μήνυμα. Υπάρχει πίεση στα κρατικά ομόλογα. Και όταν το είπα, μου είπαν ότι χρειαζόμαστε μια σαφή ένδειξη, μας είπαν, ότι θέλουμε, θα πάρουμε τα λεφτά μας. Και μέχρι τότε η πίεση θα συνεχιστεί. Θα είναι ακριβώς ο δανεισμός. Και στην ουσία έχουμε μπει σε ένα φαύλο κύκλο, από τον οποίο δυσκολευόμαστε να βγούμε. Γι' αυτό εμείς, οι πράσινοι, θέλουμε να δούμε ένα ταμείο Διάσωση ε, διάσωσης του χρέους. Πρέπει κάθε χώρα να αναλάβει μια υπεύθυνη οικονομική πολιτική. Βεβαίως, αλλά για μας, εμείς, θα καταψηφίσουμε αυτή της έκθεσης. Θα ψηφίσουμε εναντίον της έκθεσης γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι όσο καλή θα έπρεπε. Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ για την σαφή και ξεκάθαρη θέση σας, όπως συνήθως. Συνήθως αυτό, έτσι μιλάτε. Κύριε Σμιτ, είστε έτοιμος? Ευχαριστώ. Και κατόπιν ο κύριος Φόξ. Κύριε Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη που άργησα. Έγινε μια κρόαση με τον Μάριο Ντράγκη και τέθη το ίδιο ζήτημα. είναι σημαντικό όλα να πάνε με τη σειρά που πρέπει. Δεν μπορεί κανείς να, να μιλήσει για τραπεζική ένωση και να φανταστεί ότι αυτή δημιουργήθηκε. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ευρωμόλογα ή ομόλογα σταθερότητας και νάτα. Όχι. Όλα πρέπει να γίνουν με την σωστή του σειρά. Ιδάλλως δεν θα είναι καλό το αποτέλεσμα. Και όπως είπατε, η Δημοσιονομική Ένωση δεν μπορεί να ξεκινήσει με ένωση μεταβιβάσεων. Και αυτό είναι σωστό. Το θέμα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Μπορώ να συμφωνήσω για ένα ταμείο εξαγοράς του χρέους, ένα redemption fund, ε, όπως λέγεται στη Γερμανία, όπως είπαμε στη Γερμανία. Υπάρχουν διστάμενες απόψεις σε όλες τις ομάδες. Εν πάση περιπτώσει στη δική μας ομάδα υπάρχουν διστάμενες απόψεις. Δεν θα, ήταν, δεν, θα σας το πω, δεν θα σας το πω τόσο υπεραπλουστευτικά για να πω ότι ο διαχωρισμός είναι γεωγραφικός. Υπάρχουν όμως διστάμενες απόψεις και το θέμα είναι πού είναι το κράτος στο οποίο ανήκουμε και πώς το κράτος μέλος προσπάθησε να επιλύσει τα προβλήματά του ιστορικά ή και τώρα. Μελέτησα εδώ τις διάφορες προτάσεις. Πρέπει πιστεύω να τις μελετήσω κι άλλο σήμερα το βράδυ και θα γίνει μια συζήτηση μετά την συνεδρία της ομάδας μας. Κάποιες από τις προτάσεις θα τις υποστηρίξουμε, όμως δεν μπορούμε όλες. Ε, κάποιες θα τις υποστηρίξουμε έστω και διστακτικά, έστω και απρόθυμα. Αλλά πρέπει να ξέρουμε και ποια είναι και η πλειοψηφία. Η άποψη της Επιτροπής αυτής δεν νομίζω ότι ταυτίζεται με την άποψη της Επιτροπής ΕΚΟΝ. Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Όπως είπα και προηγουμένως, όπως είπε και η κυρία Τούρναν ε, που κάθεται από πίσω μου, αυτό δεν θα λύσει την κρίση στην Ευρώπη, τα ομόλογα σταθερότητας. Όμως μπορεί να ανοίξει ένα δρόμο, να είναι μια κατεύθυνση Οπότε σε αυτή την περίπτωση ίσως αύριο να πετύχουμε μια ισόρροπη προσέγγιση. Για σήμερα θα σταματήσω εδώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. ο κύριος Φόξ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να παραδεχτώ ότι μπερδεύτηκα λίγο. Γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση στην ΙΜΚΟ. Πριν από δύο εβδομάδες έγινε η ίδια συζήτηση στην Επιτροπή Και πρέπει να πω ότι δύσκολα μπορώ να σκεφτώ πώς αυτό επηρεάζει την ενιαία αγορά. Βεβαίω είναι καλό να κάνω μια συζήτηση με φύση συναδέρφου για το θέμα αυτό, αλλά δεν είμαι βέβαιο ότι αυτό θα επηρεάσει καθόλου την εσωτερική αγορά. Η ομάδα μου δεν συμφωνεί απόλυτα με το να υπάρχει μια κοινοκτημοσύνη του χρέους. Τι γίνεται η κυρία Τούρν μίλησε για τους δανούς τραπεζίτες. Αυτοί θέλουν σαφή ένδειξη ότι τα χρήματά τους τους επιστραφούν. Έχει δίκιο. Γι' αυτό ακριβώς τα κράτη που είναι καλές θετικά μπορούν να δανειστούν για 10 χρόνια. Αλλά αν έκανε δεκαετή έκδοση ομολόγων η Ελλάδα σήμερα θα πλήρωνε ε, πάνω από 1,5% που πληρώνει η Γερμανία, ίσως και πάνω από 15%. Αν ε, λοιπόν οι τραπεζίτες λένε ότι θέλουν να εξασφαλιστούν να θα πάρουν τα λεφτά τους, αυτό που εννοούν είναι ότι θέλουν να τα εγγυηθεί η Γερμανία. Αυτό εννοούν. Γιατί αυτή είναι η μοναδική εγγύηση εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει οποιοδήποτε νόημα. Τα άλλα 26 κράτη-μέλη μπορούν να γράψουν το όνομά τους, αλλά τα επιτόκια δεν θα πέσουν. Και αυτό θέτει και ένα πολύ ενδιαφέρον φιλοσοφικό ζήτημα. Γιατί πολύ συχνά στην Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε για την κοινοτική μέθοδο, αλλά όταν μιλάμε για τα ευρωομόλογα, μιλάμε για απόφαση της κυρίας Μέρκελ. Ή θα υπογράψει την επιταγή και θα λειτουργήσει το σύστημα ή δεν θα την υπογράψει και δεν θα ξεκινήσει το ευρωομόλογο. Ως Βρετανός, ξέρω ότι η χώρα μου δεν θα συμμετάσχει στα ευρωομόλογα, Θέλουμε η κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κρίση του ευρώ να επιληθεί όσο το δυνατόν ε, γρηγορότερα και θέλουμε επίσης να πάνε καλά τα μέλη της Ευρωζώνης. Η ουσία είναι όμως ότι βρισκόμαστε σε αυτό το χάλι λόγω της υπερβολικής δαπάνης και του υπερβολικού χρέους. Άρα η ιδέα ότι αν επιτρέψουμε στις υπερχρεωμένες χώρες να δανειστούν περισσότερο επειδή έχει εγγυηθεί το δανεισμό της Γερμανία η κατάσταση θα βελτιωθεί κατά την άποψή μου είναι περίεργη τουλάχιστον. Το πρόβλημα είναι πρόβλημα χρέους και δεν θα επιληθεί μέσω επιπλέον δανεισμού. Είμαι λοιπόν διατεθειμένος να επιτρέψω στα μέλη της Ευρωζώνης να δουν πώς μπορούν να λειτουργήσουν τα ομόλογα σταθερότητας, αν θεωρήσουν ότι μπορούν εν μέρει να λύσουν το πρόβλημα, ας κάνουμε μια ενδελεχή ανάλυση. Αλλά τα θεμελιώδη προβλήματα της Ευρωζώνης είναι ότι από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το ευρώ, εδώ και 12 χρόνια, η γερμανική οικονομία και η, οικονομία των κάτω χωρών και άλλες οικονομίες γίνονται ισχυρότερες, πιο αποτελεσματικές. Οι εργαζόμενοι τους εργάζονται πιο σκληρά από εργαζόμενους άλλων χωρών που δεν, η οικονομία τους δεν είναι τόσο αποδοτελική. Είναι πολύ απλό. Κάποιες χώρες δαπανούν πάρα πολύ και πληρώνουν υπερβολικά τους εργαζόμενους τους και δεν είναι ανταγωνιστικές. Η χώρα μου επί 13 χρόνια έκανε το ίδιο. Επί 13 χρόνια ε, ξοδεύαμε και δανειζόμασταν υπερβολικά. Ευτυχώς μπορέσαμε να μειώσουμε κατά ένα τέταρτο κατά 25% το νόμισμά μας για να βρούμε μια λύση. Δεν περηφανεύομαι γι' αυτό, αλλά τουλάχιστον έχουμε ένα μηχανισμό επίλυση. Αλλά υπάρχουν χώρες στην Ευρωζώνη που δεν έχουν τέτοιο μηχανισμό και δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα βοηθηθούν με περισσότερο δανεισμό. Αυτό θα το αφήσω στην κυρία Μέρκελ. Εκείνη θα αποφασίσει αν είναι διατεθειμένη να υπογράψει μια μεγάλη γερμανική επιταγή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φόξ. Σήμερα το απόγευμα όλοι μιλάμε πολύ ειλικρινά από ό,τι παρατηρώ. Θέλει κάποιος να σχολιάσει. Η κυρία Τούρναν. Θέλω να αντιδράσω, κυρία Τούρναν και μετά ο κύριος Φαμπ. το σέβομαι ε, ε, ότι κάποιοι έχουν αναλύουν τα πράγματα έτσι. Ότι η κρίση αυτή οφείλεται αποκλειστικά σε υπερβολικές δαπάνες. Αλλά για μένα αυτό είναι περιβολικά απλουστευτικό. Το επίπεδο της Ισπανίας το επίπεδο του χρέους της Ισπανίας είναι χαμηλότερο από της Γερμανίας. Η Ισπανία ήταν φτωχή πριν από μέχρι 20 χρόνια και έχει ανεβεί πάρα πολύ. Βεβαίως το παραγωγικό του μοντέλο είναι υποαμφισβήτητη ενδεχομένω. Ε, πρέπει να διαρθρώσουν την οικονομία του, να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά του. Αλλά όλα αυτά είναι μακροπρόθεσμα. Προ το παρόν, όταν υπάρχει μόνο ένα νόμισμα, ένα επιτόκιο και αν δεν διορθωθούν τα μακροοικονομικά, πού θα πάμε. Υπάρχει ένα συστημικό σκέλος εδώ, ένα συστημικό ζήτημα. Δεν είναι απλώς οι υπερβολικές δαπάνες. Βεβαίω πολλά πρέπει να αντιμετωπιστούν σε κάθε χώρα χωριστά. Αλλά αν δεν αντιμετωπίσουμε και το συστημικό σκέλος, θεωρώ ότι ε, το ευρώ θα, θα εξαφανιστεί ω νόμισμα και αυτό είναι κρίμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ηθικός κίνδυνος. Εξαρτάται πώς θα σχεδιαστεί το όλο πακέτο και τι κίνητρα θα παρασχεθούν. Θέλησα να πάρω το λόγο. Ε, ε, σέβομαι ότι η ανάλυση σας είναι διαφορετική. Θέλω όμως να πω αυτά που είπα. Ε, λοιπόν, ας ακούσουμε κι άλλες αντιδράσεις. Ο κύριος Σβάμπ, κυρία Πιετικάινεν και ο κύριος Σμιτ. Λοιπόν, ας κάνουμε μια συζήτηση, σύντομη συζήτηση από αυτού. Θα δώσω το λόγο μετά στην Υπάρχει κάποιος από την ε, ε, Κομισιόν που θέλει όχι, οπότε τα μέλη του Κοινοβουλίου εδώ έχουν ε, ελευθερία. Παρότι ο κύριος Φόξ λέει ότι δεν εμπίπτει απόλυτα στο πεδίο μας, αλλά έχουμε τουλάχιστον δικαίωμα να πούμε ένα λόγο περί αυτού. κύριος Φαμπ, η κυρία Πιέτη Κάινεν και ο κύριος Σμιτ και άλλοι. Και ο κύριος Φόξ. Έχετε δικαίωμα κι εσείς να ακουστείτε. Μην μακρηγορήσει κανένας, αλλά έχουμε χρόνο για κάποιους ομιλητές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση ε, έχει ως εξής. Ε, μιλάμε στην Επιτροπή για αυτό το θέμα, ούτως ή άλλως και πρέπει να το κάνουμε επικοδομητικό το διάλογο. Δεύτερον, δεν έχει να κάνει τόσο με το τι θέλουμε. Ε, δεν είναι πάντοτε αυτή η κατάλληλη συνταγή να πάμε ε, πάντοτε προς τη λύση για τις ε, τράπεζες, για παράδειγμα. Δεν έχουν ασφαλή τράπεζες και δεν υπάρχει ασφάλεια σε αυτόν τον κόσμο και γι' αυτό είναι τόσο πολύπλοκο το θέμα. Επίσης, υπάρχουν και τα συστημα... οι συστημικοί κίνδυνοι Υπάρχει αυτό το θέμα της κοινή ευθύνη. Άρα εμείς ως ε- ε- Ευρωπαίοι, γνωρίζοντας ότι είναι απαραίτητη η αλληλεγγύη και μόνο έτσι μπορούμε να κερδίσουμε στο μέλλον, προχωράμε με αυτό το, σε αυτό το δρόμο, όμως υπό τον όρο ότι όλοι θα κάνουν εξοικονόμηση, ότι θα μπορέσουν ε, να αναγνωρίσουν αυτό τον ηθικό κίνδυνο ενός, μιας κοινοκτημοσύνης ενδεχομένως του χρέους. Επίσης για το Tupac δεν είχε ε, την πλειοψηφία και όλοι λέγαμε ε, ότι πρέπει να το υπερψηφίσουμε παρόλο που δεν είχαμε την αρμοδιότητα. Άρα, σε αυτά τα δύσκολα ζητήματα το Κοινοβούλιο πρέπει να δείχνει η αλληλεγγύη παρόλο που οι σοσιαλιστές ε, μας εξεπατούν σε αυτό και γι' αυτό σε αυτή την Επιτροπή βλέπουμε πόσο θετική είναι η προσέγγιση. Απ' την άλλη, ε, γενικά επί της αρχής συμφωνούμε, όμως ε, όλοι λέμε ότι πρέπει στο μέλλον, για να υπάρχει κοινό ε, μέλλον, να υπάρχει μια κοινή ευθύνη, αλλά αυτό πολιτικά και νομικά να γίνει σωστά, ώστε να μπορούν και οι δύο πλευρές να προχωρήσουν σωστά και γι' αυτό πρέπει να εξετάσουμε το συμβιβασμό, να δούμε, ε, να εξασφαλίσουμε ε, πώς μπορεί κάθε πλευρά να προσεγγίσει την άλλη έτσι ώστε να υπάρχει μια ρύθμιση που στο τέλος θα οδηγήσει σε λύση σωστή και για τις δύο πλευρές. Και είναι πολύ καλό που συζητούμε αυτό το θέμα κύριε Πρόεδρε, όπως έγινε και στην ΕΚΟΝ και ε, πραγματικά μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια επικοδομητική λύση. Ωραία. Η κυρία να έχει το λόγο. Δεν, Δεν ξέρω πόσο ωφελεί να παρέμβει κανείς σε αυτή τη συζήτηση, αλλά προκλήθηκα και θα απαντήσω. Και μετά από τι ε, είπε ο Σφάμπ. Μπερδεύομαι λίγο καμιά φορά όταν ακούω ότι μιλάμε, όταν μας ακούω να μιλάμε για ευρωμόλογα. Μιλάμε για αυτά τα χρεόγραφα του υφιστάμενου χρέους. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Αλλά εξ όσων αντιλαμβάνομαι εγώ, όταν μιλάμε για τα ομόλογα σταθερότητας, μιλάμε για κάποιο μελλοντικό στοιχείο που θα σταθεροποιήσει το ευρώ και την ευρωπαϊκή αγορά υπό την έννοια μπορεί να είναι θέμα εσωτερικής αγοράς, γιατί δεν μπορεί κανείς να έχει καλή εσωτερική αγορά αν δεν υπάρχει σταθερότητα. Επίσης για μένα είναι ένα θέμα θέμα αυτή η λιτότητα ή η, η κοινη ανάληψη ευθύνης. Δεν μπορεί να υπάρχει το ένα χωρίς το άλλο. Και για μένα υπάρχει μια αλληλουχία και αυτό δεν είναι πιο δύσκολα από ό,τι κάνουμε στην ιδιωτική μας ζωή. Δεν πρέπει να εγγυόμαστε ε, τα χρέη κάποιου αν δεν έχουμε κάποια εξασφάλιση ή αν δεν γνωρίζουμε ότι ο άλλος θα μπορεί να αποπληρώσει το χρέος του. Αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα για την Ευρώπη. Εγώ είμαι πολύ υπέρ των ομολόγων σταθερότητας κάποια στιγμή στο μέλλον όταν πλέον πολλά πράγματα θα έχουν μπει στη θέση τους. Και βεβαίως το Ταμείο Εξαγοράς του Χρέους θα είναι μια καλή λύση αλλά υπάρχουν μια ολόκληρη σειρά αποζητήματα για το πώς θα λειτουργήσει, ποιος θα παρέχει τις εγγυήσει. Δεν είμαι ε, σίγουρη ότι οι Φιλανδοί και οι Γερμανοί θα είναι πρόθυμοι να το κάνουν. Επίσης, το άλλο θέμα επί του οποίου θα ήθελα, το οποίο θα ήθελα να υπογραμμίσουμε με είναι ότι η δομή των red chips και των blue chips θα είναι καλή ιδέα. Ιδάλλως τα spread θα είναι πάρα πολύ υψηλά. Υπάρχουν δηλαδή τα ομόλογα σταθερότητας με διαβάθμιση ΑΑ στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και υπάρχουν και αυτά της κατηγορίας Β που προσπαθούν να φτάσουν εκεί. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σμιτ και μετά ο κύριος Κορέα Ντεκάμπος, μετά από όλους τους ομιλητές. Ο κύριος Φόξ και εγώ βρισκόμαστε εκτός σχήματος. Γι' αυτό ίσως δεν θα έπρεπε να συμμετέχουμε έχουμε καν σε αυτή τη λογομαχία. Εάν όμως τα ομόλογα σταθερότητα σχετίζονται με το ευρώ, και περί τίνος ε, πρόκειται, γιατί το ευρώ σχετίζεται με την εσωτερική αγορά, με την ενιαία αγορά. Και από βρετανικής πλευράς θα πρέπει να κρατήσουμε ένα ενιαίο σταθερό πλαίσιο για την ε, αγορά, για την εσωτερική αγορά. Εάν λοιπόν το ευρώ αντιμετωπίζει προβλήματα, και αυτό ήδη ελέγχθη από τη Βρετανική πλευρά τους Βρετανούς Υπουργούς και συνάντησα και έναν δύο ώρες πριν. Αυτό θα επηρεάσει τη Σουηδία και τη Βρετανία. Υπάρχει δηλαδή η αιτιώδη συνάφεια εδώ. Εγώ προέρχομαι από μία χώρα όπου πάντα προσπαθούσαμε να επιλύσουμε τα προβλήματά μας σε σχέση με την υποτίμηση. Και αυτό τι σήμαινε, ότι γίναμε όλα ένα πιο φτωχοί, προσπαθήσαμε να περισσώσουμε το νόμισμά μας και μόνον. Άρα δεν είναι αυτός ο τρόπος. Αν όλες οι χώρες υποτιμήσουν, και δεν μπορείτε να το προτείνετε αυτό, θα ήταν καταστροφή. Χρειαζόμαστε δημοσιονομική εξυγίανση και διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Και όπως είπε και ο κύριος Σφαμπ, το χρειαζόμαστε με μια συγκεκριμένη τάξη και ιεράρχηση. Γι' αυτό απασχολεί και τη Γερμανία. Θα πρέπει να είμαστε περήφανοι για τη Γερμανία. Γιατί όλο και κάτι καταβάλλεται. Εμείς δεν καταβάλουμε τίποτα. Και αυτό συζητιέται και στη Φιλανδία. Βρέθηκα εκεί ε, μερικές εβδομάδες πριν. Δεν δείτε τι γίνεται τι γίνεται με τη Σουηδία και τη Φιλανδία. Τι κάνουν ε, οι βαλτικές χώρες, ας πούμε, δεν καταβάλουν τίποτα, όμως θα καταφέρνουν εξίσου καλά ε, με εμάς. Περί αυτού πρόκειται, περί αλληλεγγύης και αυτό θα πρέπει να αφορά και την Μεγάλη Βρετανία και τη Δανία. Η κυρία Φερχάιεν. Να συζητήσω ένα θέμα που πρέπει να διευκρινιστεί. Δεν είναι το ευρωομόλογο η λύση του προβλήματος της κρίσης είναι το ε, περιθώριο, το πλαίσιο το οποίο συζητάμε και είναι απαραίτητο. Θα ήθελα περισσότερο η έκθεση να μιλά για τις ε, προϋποθέσεις πλαίσιο, με ποια μορφή θα έχουν, ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις, έτσι ώστε οι μικρομισές επιχειρήσεις να μην πλήττονται. Γιατί οι προϋποθέσεις πλαίσιο που είναι απαραίτητες για να λειτουργήσουν τα ομόλογα σταθερότητας είναι αυτό που αναφέρεται συνεχώς ε, στο κείμενο. Αυτό είναι που θα μας πάει μπροστά και αυτό ε, αναφέρεται συνεχώς στο κείμενο ότι τα ευρωομόλογα σταθερότητας πρέπει να είναι μόνο το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας η οποία θα οδηγεί σε περισσότερη σταθερότητα, ευθύνη οικονομική, χρηματοοικονομική και ε, για μια, το αποτέλεσμα μιας ε, διαδικασίας ε, ε στην οποία, η οποία αν δεν υπάρχει δεν θα έχουν καμία ε, απο, δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα τα ομόλογα σταθερότητας. Οι Γερμανοί συνεχώς μπαίνουν στο προσκήνιο, όμως θα πρέπει όλοι να κάνουν το δικό τους μερίδιο έτσι ώστε στο διηνεκές να είναι ε, σίγουρα τα ομόλογα αυτά. Έχουμε λοιπόν ε, να δούμε, πρέπει να δούμε και πόσο μπορεί να διαρκέσει μια οικονομία. Δηλαδή πριν την εισαγωγή των ε, ομολόγων σταθερότητας πρέπει να δούμε αν πληρούνται οι προϋποθέσεις και αυτό σημαίνει ότι διαρθρωτικά θα πρέπει να δούμε και τον δρόμο που θα ακολουθήσουμε προς μεγαλύτερη αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη ε, δεν είναι κάτι, ένας δρόμος στον οποίο διανύει κανείς μόνος του. Πρέπει όλοι να κάνουν το μερίδιό τους, να βάλουν το λιθαράκι τους. Και μόνο έτσι ε, θα μπορέσουμε να δούμε πώς θα κάνουμε τα ομόλογα σταθερότητα την αρχή μιας διαδικασίας. Η ίδια όμως η διαδικασία είναι που θα ε, διατηρήσει την ισχύ της οικονομίας μας και αυτά τα ομόλογα θα μπορούν να είναι μόνο μία κρίσιμη μάσα που θα υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία έτσι ώστε να καταλήξουμε σε αυτό που ξεκάθαρα δείχνει η έκθεση. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πραγματικά διαφωτιστική η συζήτηση. Ε, ζητώ συγγνώμη που κράτησε τόσο η συζήτηση, αλλάξιζε τον κόπο νομίζω. Η κυρία Ρικόινεν, συγγνώμη, εσείς θα μιλήσετε τελευταία. Απλώς θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ στη χώρα μου, γιατί πολλοί αναφέρθηκαν σε αυτήν. Ο κύριος ε, Κορέιρα και η κυρία Τούρουνεν προσπάθησαν να υποστηρίξουν τη χώρα μου. Θεωρώ ότι ορισμένα θέματα είναι σημαντικά εάν θέλουμε να επιλύσουμε το ζήτημα του ευρώ και του χρέους. Αυτό είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί όλους. Και επειδή θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί, όπως και η κυρία Τουρούνεν, θα πρέπει να ξέρετε ότι αυτά που λέτε για τη χώρα μου δεν αντικατοπτρίζουν την αλήθεια. γιατί θα πρέπει να μην παρατείνουμε την αγωνία του ασθενούς, να μην τον έχουμε στην εντατική. Πρόκειται για μία άδικη αγωνία για τους Ισπανούς και γι' αυτό θα πρέπει να αλλάξουμε τις αντιλήψεις. Γιατί μιλάμε για βασικές έννοιες φερεγγιότητα, σπουδή και λιτότητα. Εμείς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση με όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Και αυτό είναι ύψης της σημασίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για μια βαριά πέτρα που μας πιέζει και δυστυχώς δεν έχουν αναλυφθεί κοινέ αποφάσεις. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να σταματήσουμε την οδό, στην οδό των αμφιβολιών και να λάβουμε δραστικές αποφάσεις. Ωραία. Δίνω τώρα το λόγο και πάλι στον εισηγητή για ένα σύντομο ε, καλακταλεκτικό σχόλιο. Ευχαριστώ άκρος ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση. Εγώ δεν συμμετείχα γιατί έθεσα ερωτήματα στην αρχή και μίλησα για ένα διαδικαστικό πλαίσιο, όμως θα ήθελα τώρα να πω ε, μερικά, να θίξω ορισμένα θέματα. Κινηθήκαμε μέχρι εκεί που μπορούσαμε, γιατί υπήρχαν αντιγνωμίες και πολλοί συνάδελφοι είναι επιφυλακτικοί σε σχέση με την υποστήριξη προτάσεων. και εμείς έχουμε εκφράσει πολλές επιφυλάξεις, ιδιαίτερα σε μία πρόταση συμβεβασμού που αποσύραμε για λόγους έλλειψης συνένεσης που βασιζόταν στο Τούπακ στα δύο νομοθετήματα. Άρα η σκιώδης ήταν επιφυλακτική. και ευθυγραμμιστήκαμε κι εμείς. Θα ήθελα να πω ότι για μας αυτό αποτελεί θυσία, μεγάλη θυσία. Οι λύσεις και τα σχόλια που αφορούν ορισμένες χώρες ε, θα πρέπει να μην είναι μανιχαϊστικής φύσης, δηλαδή οι καλοί και οι κακοί, ποιοι εργάστηκαν και ποιοι δεν εργάστηκαν. Αυτό δεν τιμά την Ευρώπη. Γιατί δεν υπάρχει και αληθοφάνεια. Το 75% των εμπορικών συναλλαγών διενεργούνται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για ένα 75% και αν υπάρχουν χώρες με πλεόνασμα, έχουν πλεόνασμα διότι άλλες έχουν έλλειμμα. Είναι σαφέστατο αυτό, δεν υπάρχει κανένας άλλος μαθηματικός νόμος ή κανόνας ή υπολογισμός. Δεν πρέπει λοιπόν να υπάρχει αυτή η μανιχαϊστική προσέγγιση. Δεν είναι επικοδομητική αυτή η προσέγγιση. Το παρόν διαφέρει από το παρελθόν. Και βεβαίως πολλές χώρες ε, πληρώνουν πολύ ακριβά το τίμημα λαθών του παρελθόντος. Στη χώρα μου, δυστυχώς, το Συνταγματικό Δικαστήριο ε, έλαβε συγκεκριμένες αποφάσεις. Μειώθηκαν οι μισθοί, ε, μειώθηκαν οι συντάξεις για να φτάσουμε σε δύο δις εξοικονομήσεις και θα το καταφέρουμε. Να μην έχετε καμία αμφιβολία. Με μεγάλες θυσίες θα, θα τα καταφέρουμε. όπως και το κάναμε στην περίοδο της δεκαετίας του 80, διότι τότε έπεσε το έλλειμμά μας από 7% σε 2%. Τότε ε, η Ισπανία είχε μεγάλο πλεόνασμα. Άρα δεν δεχόμαστε τα μανιχαϊστικά σχόλια που ακούγονται για την κατάσταση και την αντιμετώπιση της. Γιατί οι λογαριασμοί δεν σημαίνουν μόνο έλλειμμα και δημόσιο χρέος. Υπάρχει και το λανθάνον χρέος που αφορά το ασφαλιστικό. Και υπάρχουν χώρες που έχουν λανθάνων χρέος που είναι το διπλό του ΑΕΠ τους. Απλώς δεν θέλω να πω ποιες είναι αυτές οι χώρες. Ξέρουμε όμως ποιες είναι. Άρα κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν θα πιω από αυτό το νερό, όπως λένε και τα Ευαγγέλια. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν θα πιω από αυτή την πηγή. Δεν πρόκειται για μια θαυματουργή λύση, δεν πρόκειται για ένα silver bullet. Εάν όμως αποστείλουμε ένα αρνητικό μήνυμα για την σκοπιμότητα ή βιωσιμότητα των ε, ομολόγων αυτών, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο πρέπει να ε, εισαχθούν αυτά τα ομόλογα σταθερότητας, να δούμε τη σκοπιμότητα υπάρχει ή δεν υπάρχει. Υπάρχουν αρνητικά στοιχεία. Έχουμε να διανύσουμε πολύ μεγάλο δρόμο και βρισκόμαστε στην απαρχή μιας διαδικασίας, κάτι το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει αύριο στην ψηφοφορία μας υποβάλλατε τους συμβιβασμούς. Υπάρχουν και κάποιες τροπο, ε, προφορικές τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. Θα δούμε το αποτέλεσμα αύριο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Οπότε πλέον, επειδή έχουμε και κάποια καθυστέρηση, ε, θα ζητήσω συγγνώμη από την εισηγητή, τη συντάκτρια της γνωμοδότησης και θα περάσουμε στην πρόταση κανονισμού ε, για τις υπηρεσίες εδάφους αριλημένες της ε, Ένωσης. Έχουμε και τους σκιόδης, Σαλτιμόσα, Παρπάνοβα, κυρία Ρούλα και έναν σκιώδη που είναι απόν. Υπάρχει και εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βεβαίως. Ωραία. Και η κυρία Μέα, λοιπόν, από την Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση MOVE, η οποία και αυτή θα συμμετέχει στη συζήτηση. Ας ακούσουμε λοιπόν την ε, εισηγήτρια την κυρία Γκάλ Πέλτς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τους και όλους εισηγητές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επικοδομηνική συνεργασία τους στο σχέδιο αυτό γνωμοδότησης. Χαίρομαι πολύ που μπορεί το Κοινοβούλιο να ε, στείλει ένα σαφές ε, μήνυμα υποστηρίζοντας το θέμα της ισόρροπης απελευθέρωσης των ε, υπηρεσιών εδάφους στους Στο, σε στο σύντομο διάστημα που ασχολήθηκα προσπάθησα να συζητήσω ο, όλες τις πλευρές του θέματος. Το λεπτότερο θέμα είναι εάν χρειάζεται υπεραιτέρω απελευθέρωση. Επειδή η οδηγία ε, ξεκίνησε ως μια προσπάθεια πολλών βημάτων έπρεπε να δούμε αν θα υπάρξει όφελος από την απελευθέρωση της αγοράς υπηρεσιών εδάφους, αν θα υπάρχει δηλαδή προστιθέμενη αξία και επίτευξη των στόχων του κειμένου. Αυτό μπόρεσε να γίνει με την αύξηση του αριθμού των ε, προμηθευτών, των τρίτων προμηθευτών και θα οδηγούσε στην τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής με επιπλέον κανόνες σε περιπτώσεις που ε, είναι μεγάλη η αγορά του αεροδρομίου. Χρειάζεται όμως να υπάρξει μια νέα ανεξάρτητη ανάλυση επιπτώσεων πριν προχωρήσουμε στην απελευθέρωση στην πρόταση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυξάνει την υποχρέωση του ελάχιστου αριθμού ε, τρί, ε, παρόχων, τρίτων παρόχων σε υπηρεσίες εδάφους από δύο σε τρεις παρόχους, ένα αεροδρόμιο, που ε, θα έχει πάνω από 5 εκατομμύρια επιβάτες και, και με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει μεγαλύτερη επιλογή και θα μπορέσει να υπάρξει καλύτερη, καλύτερη ποιότητα ε, υπηρεσιών εδάφους. Όπως είπα και στην προηγούμενη συνεδρία της Επιτροπής, καθώς ε, παρουσίαζα το σχέδιο γνωμοδότησής μου, πιστεύω ότι το άνοιγμα πρέπει να γίνει με τρόπο ισόρροπο. Έχουμε προετοιμάσει συμβαστικές τροπολογίες από αυτού και με βάση αυτή τα αεροδρόμια που έχουν ετήσια ε, αριθμό επιβατών πάνω από 5 εκατομμύρια ή 100.000 τόνοι φορτίου τα τελευταία τρία χρόνια, η Επιτροπή θα θεωρήσει ότι υπάρχει λόγος αύξησης του αριθμού των παρόχων υπηρεσιών εδάφους από 2 σε 3, σε 3 και αυτό θα υποβληθεί σε κάποια εθνική εποπτική αρχή, η οποία ως ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή θα αποφασίσει με βάση τις ιδιαιτερότητες ανάλογα με την κάθε κατηγορία υπηρεσιών εδάφους με διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις. Το δεύτερο πακέτο συμβιβασμών ε, αφορά τα πρότυπα ποιότητας για τον ανεφοδιασμό και το χειρισμό των αποσκευών μέχρι και τις διαδικασίες check-in. Προσπάθησα να βρω συμβιβασμό με την εισαγωγή ενός νέου άρθρου που διευκρινίζει τι είναι αυτά τα ε, πρότυπα ποιότητας. Είμαι υπέρ της εισαγωγής ελάχιστων προτύπων που βελτιώνουν τις υπηρεσίες και θα βοηθήσουν τη λειτουργία των αεροδρομίων. Είναι σημαντικό τα ελάχιστα πρότυπα να σέβονται τους ε, κανονισμούς, τις απαιτήσεις ασφάλειας, ανάλογα με τους κανονισμούς και τους κοινούς κανόνες στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας. Κατόπιν, εισάγω την υποχρέωση για τους παρόχους υπηρεσιών εδάφους να δημιουργήσουν ένα σύστημα ασφαλούς διαχείρισης όπου θα επιβάλλονται τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητος. Επιπλέον, οι αρχές λειτουργίας του ε, αεροδρομίου έχουν την υποχρέωση να επιβάλλουν αυτά τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας. Έχουμε συζητήσει και άλλα θέματα, όμως νομίζω ότι ε, κοινωνικά θέματα, αλλά αυτο νομίζω είναι στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Απασχόλησης. Ε, ένα άλλο θέμα είναι η, η ανάθεση των υπηρεσιών σε τρίτους. Η ευθύνη αυτών των υπηρεσιών θα υπόκειται σε ελέγχους με σκοπό την εξασφάλιση και του δικαίου ανταγωνισμού. Και εδώ υπάρχει συμβιβαστική πρόταση. Τέλος, θα πρέπει να παρέχεται ένα επαρκές επίπεδο εκπαίδευσης σε όλο το προσωπικό και όχι μόνο στο προσωπικό ασφαλείας των οργανισμών ε, παροχή υπηρεσιών εδάφους. Θεωρούμε ότι όλα αυτά είναι σε όφελος όλων των επιβατών των, ε, και του προσωπικού. Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχουν μονοπωλιακές συνθήκες και ότι θα υπάρξουν ξεκάθαροι κανόνες για τους χρήστες. Για μία ακόμα φορά θέλω να ευχαριστήσω για τη δουλειά τους τους σκιώδες εισηγητές, τη γραμματεία της Επιτροπής, όπως και όλους όσοι ασχολήθηκαν με το δύσκολο και σύνθετο αυτό ζήτημα. Θεωρώ ότι οι συμβιβαστικές προτάσεις είναι καλές και προσθέτουμε προς τη θέμενη αξία στους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Πέλτς. Øh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας στον εισηγητή ότι είμαι ευγνώμων για αυτή την εξαίρετη συνεργασία επί της προτάσεως αυτής. Είναι επικοδομητική και πραγματικά είμαι σίγουρη ότι είναι ένα αποτέλεσμα πολύ καλό με βάση και τις συμβαστικές ε, τροπολογίες. Ε, για την ομάδα μας ε, να πω ότι η Κομισιόν ξεκίνησε το δρόμο αυτό Όμω, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για τα κράτη-μέλη και όχι κάτι που τους επιβάλλεται και νομίζω ότι έχει, βρίσκεται στη σωστό δρόμο ε, η πρόταση. Θα πρέπει να υπάρχουν τα ελάχιστα στάνταρ, οι ελάχιστε προδιαγραφέ για τις υπηρεσίες ε, στα αεροδρόμια και για τις υπηρεσίες εδάφου. Τέλος, να πω ότι ήταν σημαντικό για μας ε, να βρούμε και μια σωστή ισορροπία ως προς την προστασία των εργαζομένων στα αεροδρόμια. Και νομίζω ότι ο συμβιβασμός ε, ήταν πολύ ικανοποιητικό συνολικά. Λοιπόν, είμαστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα και νομίζω ότι ε, μόλις ψηφίσουμε αύριο η Επιτροπή Μεταφορών θα χρησιμοποιήσει τις εξαίρετες προτάσεις μας. Ευχαριστώ πολύ για την καλή σας συνεργασία. Ευχαριστούμε την κυρία Σαρλαμέτσα και την κυρία Παρβάνοβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υποστηρίζω την προσέγγιση του εισηγη... της εισηγητρίας. Θεωρώ ότι έχει φτιάξει μια ισορροπημένη και συνολικά ε, καλή ε, γνωμοδότηση. Θα Μάλλον περιμένω ότι η Επιτροπή μας ε, θα παρουσιάσει την λιγότερο αμφισβητούμενη γνωμοδότηση σε σχέση πούμε, με την Επιτροπή Έργαση Employment. Υπάρχουν πολύ σημαντικά θέματα όπως οι σωστές ε, ε, η σωστή εργασία για τους εργαζομένους, τα ελάχιστα στάνταρ, η σωστή εφαρμογή. Υποστηρίζω τη σταδιακό άνοιγμα των υπηρεσιών ε, εδάφους, ε, σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν, αυτό θα πρέπει να γίνει μετά από την ρύθμιση, αφού δηλαδή η πρόταση εφαρμοστεί από τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό ε, δεν υποστηρίζουμε τις τροπολογίες που ζητούν για μεγαλύτερο άνοιγμα, μιλούν για μεγαλύτερο άνοιγμα της αγοράς και ε, υποστηρίζουν την δυσανάλογη κοινωνική προστασία των ε, εργαζομένων. Οι συμβιβαστικές τροπολογίες είναι μια λύση που ικανοποιεί όλους νομίζουμε. Θα τις υποστηρίξουμε και αυτή την προσέγγιση θα την υποστηρίξει και η Αρμόδια Επιτροπή αν έχουμε καλή τύχη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Να δούμε ποιος άλλος είναι η κυρία Ρούιλε. Θα ήθελα κι εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια καταρχάς ε, για την έκθεση της. Θεωρώ ότι η έκθεσή της ήταν μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής γιατί μιλάει για την απέτηση για στάνταρ ποιότητας ε, και ασφάλειας και αυτό είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη. Η έκθεση επίσης τελικά ταιριάζει με την πρόταση ε, της Κομισιόν όσον αφορά στο άνοιγμα των αγορών. Θεωρώ ότι ήταν καλό που είχαμε ε, συμβιβασμό να μην είναι δηλαδή ε, υποχρεωτικό το άνοιγμα, αλλά να υπάρχει δυνατότητα ανοίγματος της αγοράς. Είναι ο σωστός δρόμος και νομίζω ότι η πρότασή μου να υποσύρει η Κομισιόν την πρότασή της ε, αρχικά διαψεύστηκε, υπήρχε μια πολύ καλή συνεργασία και τελικά είχαμε μια εξαίρετη ε, έκθεση. Πραγματικά ε, χρησιμοποίησαμε την ευκαιρία ε, για να γίνει μια καλή αναθεώρηση της πρότασης. Ευχαριστούμε την κυρία Ρούλε. Καλωσορίζω τον Τόμας Μαν που ήρθε μαζί μας σήμερα το απόγευμα και νομίζω ότι είναι και ο εισηγητής για την Επιτροπή Εργασίας για αυτό το θέμα. Ε, σας ε, καλώ λοιπόν να κάνετε ένα σχόλιο προσκεκλημένο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, χαίρομαι που βρίσκομαι σε αυτή την επιτροπή γιατί δεν είμαι, είναι πολύ μακριά από τις ιδέες που ε, τώρα εμείς υποστηρίξαμε στην Επιτροπή Απασχόλησης. Έχω κάνει μια έκθεση για αυτήν την Επιτροπή Απασχόλησης και είδαμε ότι καλό είναι να μην, παλευ... να μην ε, μαλώνουμε, αλλά τελικά να δούμε ποια είναι τα πεδία που μας ενδιαφέρουν και να βρούμε ένα καλό συμβιβασμό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε ότι δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικό το άναγμα. Το αναφέρει και η κυρία ε, Ρούλε. Το συζητήσαμε με τον Πατ Πολ και με άλλους ε, για το πώς θέλουμε να υπάρχει σταθερότητα και αυτό είναι ένα καλό μήνυμα. Σε αυτό τον τομέα συμφωνούμε. Δεύτερο η παρατήρηση που θεωρώ σημαντική. Σωστά αναφέρατε κυρία εισηγήτρια ότι μια πλήρης απελευθέρωση θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη αστάθεια. Είναι πολύ σωστό. Θα μπορούσαν να δημιουργηθούν αλληγοπόλια και θα έμεναν λιγότερες ε, επιχειρήσεις στον κλάδο. Θα ήταν αυτές οι οποίες ε, θα είχαν εξαγοράσει για να ε, ε, πάρουν την αγορά, αλλά δεν θα είχαν ε, πληρώσει αρκετά. Και αυτό θα ήταν ένα πολύ ανησυχητικό μήνυμα, γιατί θα ήταν πολύ επισφαλής η όρη εργασίας των εργαζομένων. Επίσης, οι επιβάτες θα ήταν ανασφαλείς για το πώς θα παρέχονταν αυτές οι οι υπηρεσίες. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει μια σωστή κατεύθυνση και να υπάρχει το θέμα της ποιότητας. Ευχαριστώ λοιπόν ε, και την εισηγήτρια για τα ελάχιστα ε, στάνταρ, τις προδιαγραφές που ανέφερε. Εγώ ε, ως εισηγητής της Επιτροπής Απασχόλησης στην έκθεσή μου συμπεριέλαβα το γεγονός ότι χρειαζόμαστε μία βασική ασφάλεια και ε, ποιότητα και αυτό σημαίνει φυσικά ότι και οι απασχολούμενοι θα πληρώνονται διαφορετικά από ό,τι τώρα. Και άλλος ένας τομέας που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικός είναι ε, να υπάρχει πάντοτε μια συνεχής κατάρτιση και εκπαίδευση. Ε, το να λέει η Κομισιόν ότι μέσα σε δύο μέρες κανείς έχει μάθει το θέμα, θεωρώ ότι είναι ε, μη ρεαλιστικό. Είναι πολύ διαφορετικά τα αεροδρόμια μεταξύ τους. Εγώ δεν έκανα μια έκθεση για τη Γερμανία, ε, όντως Γερμανός. Έκανα μια έκθεση για τα διαφορετικά αεροδρόμια που υπάρχουν, γιατί κάποια πράγματα λειτουργούν σε κάποια αεροδρόμια και κάποια δεν λειτουργούν σε άλλα. Υπάρχει μια σειρά παρόχων ε, ε, έχουμε συχνά ε, μία-δύο ώρες καθυστερήσεις όταν ε, το αεροδρόμιο δεν είναι σωστά διαρθρωμένο. Όταν όμως είναι σωστά διαρθρωμένο όλα πάνε πολύ γρήγορα. Πρέπει να έχουμε λοιπόν ίσες ευκαιρίες και όλοι να έχουν σωστή ποιότητα και σωστή αμοιβή. Νομίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να υπερψηφίσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες γιατί ελπίζω ότι με την έκθεσή σας θα αλλάξουν τα πρόγματα ε, στην Επιτροπή Μεταφορών. Να πω και κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε. Ε, υπόθηκε πολλές φορές ότι δεν θέλουμε κανονισμό, γιατί θεωρούμε ότι οι υπηρεσίες εδάφους είναι ένα κομμάτι ε, του γενικότερου πακέτου αεροδρομίου, ε, που παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Είμαστε έτοιμοι να πούμε ότι δεν θέλουμε κανέναν κανονισμό, αλλά θέλουμε μια οδηγία για τις ε, ιερομοδιότητες των κρατών μελών, αντί να έχουμε έναν κανονισμό, ο οποίος θα είναι ε, ένας για όλα τα κράτη-μέλη. Ε, ευχαριστώ τον Πρόεδρο λοιπόν και την εισηγήτρια για αυτή την πολύ παραγωγική συζήτηση και την σωστή πρόταση που έχει διατυπωθεί, διατυπωθεί από αυτή την Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο? Όχι. Ε, ας, δώσουμε τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την κυρία Μέγερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ στην εισηγήτρια για την εξαιρετική δουλειά που έκανε. η δουλειά που απαιτεί ειδικέ γνώσεις και συμβιβασμούς, πράγμα που δεν είναι πάντα εύκολο. Θα ήθελα να κάνω τέσσερις παρατηρήσεις. Πρώτον, όσον αφορά τις συνθήκες ανοίγματο της αγοράς. Γνωρίζετε τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία διαφέρει από τη θέση του συμβιβασμού που προτείνεται εδώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι ο ελάχιστος αριθμός παρόχων υπηρεσιών πρέπει να είναι τρεις Βεβαίω, είναι δυνατόν μεγαλύτερο άνοιγμα και κάθε κράτο μέλο, ανάλογα με τις ιδιαίτερότητε του μπορεί να καθορίσει εάν χρειάζονται περισσότεροι πάροχοι υπηρεσιών για κάποιες κατηγορίες. Είναι πολύ πρόσδεκτο το γεγονός ότι η Επιτροπή σας δεν θεωρεί τις ε, τροπολογίες, τις αυτοβοήθειες και τις ε, ανάθεση σε τρίτους. Αυτή τη στιγμή, κάποια στιγμή φοβηθήκαμε ότι θα επέλθουν αλλαγές που θα επηρέαζε την ε, αγορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επόμενο σημείο αφορά τις τροπολογίες που αφορούν τη μεταφορά προσωπικού. Ο συνδυασμός των τροπολογιών όπως έγιναν, 57 και 60, μας φάνηκε ότι δεν ήταν ισόρροπος. Επιπλέον πρέπει να επενθυμίσουμε ότι οι αγορές στις οποίες υπάρχουν περιορισμοί πρόσβασης είναι συγκεκριμένες και για τις αγορές αυτές η επιλογή των παρόχων υπηρεσιών θα γίνεται κάθε επταετία μέσω ε, υποβολής προτάσεων. Άρα η σταθερότητα θα υπάρχει για τα επτά χρόνια οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν κίνητρο να εξοικονομήσουν. Και γι' αυτό οι διατάξεις που προτείνει η Κομισιόν αφορούν τις κλειστές αγορές, τους κλειστούς διαγωνισμούς. Επιπλέον, το να πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να κάνουν μεταφορά προσωπικού θα είναι σε βάρος της ευρωπαϊκής αγοράς λόγω του κόστους και των εμποδίων εισόδου. Και αυτό αντιβαίνει στην αρχή της επικουρικότητας που, αφορά, που αφήνεται στα κράτη-μέλη το θέμα της ε, κοινωνικής στήριξης. Επίσης υπάρχει το θέμα ε, των εγκρίσεων που δεν θέλησε να στηρίξει το Συμβούλιο και το θέμα των ελάχιστων προτύπων ποιότητας. Τέλος, όσον αφορά τις παρεκκλήσεις για το άνοιγμα της, από το άνοιγμα της αγοράς, άρθρο 14, θέλαμε δύο πράγματα να υπενθυμίσουμε. Πρώτον, ότι το άρθρο 14 είναι σημαντικό, δεδομένου ότι επιτρέπει την περίπτωση εξαιρέσεων όταν υπάρχει έλλειψη χώρου σε ένα αεροδρόμιο και δεν επιτρέπει το άνοιγμα της αγοράς. Δεύτερον, ότι είναι επικίνδυνο τώρα να γίνουν τροποποίησεις ουσίας, το άρθρο 14. Το άρθρο αυτό έχει λειτουργήσει στην υφιστάμενη οδηγία, έχει αποδείξει την αξία του και έχει σημασία να διατηρηθεί. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για μία ακόμα φορά θέλω να σας ευχαριστήσω εσάς, την ε, Επιτροπή ΙΜΚΟ, για την σοβαρή και σε βάθος δουλειά που κάνατε για ένα θέμα που μας είναι προσφυλές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια σαφή επεξήγηση και για την θετική ανταπόκριση στις προτάσεις μας. Η κυρία Κέλπελ θέλει κάτι να πει καταληκτικά, εντάχει. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ανταπόκρισή σας και θεωρώ ότι η πρόταση αυτή αφορά διάφορους εμπλεκόμενους φορείς, διαπραγματευτήκαμε τα μείζωνα ζητήματα και εκεί όπου υπήρχαν ερωτηματικά. Στη γνωμοδότηση αυτή προσπαθήσαμε να φτάσουμε σε μία ισορροπημένη πρόταση και συμφωνούμε και στους συμβιβασμούς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Κιώδης και τη Γραμματεία, καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συνεργασία τους σε, αυτή την, σε αυτό το σχέδιο ονομοδότησης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την εργασία σας. Θα ψηφίσουμε αύριο το πρωί για την έκθεση αυτή. Τελική γνωμοδότηση για σήμερα είναι το σχέδιο γνωμοδότησης Κοφεράτη σχετικά με μια ατζέντα για επαρκής ασφαλής και βιώσιμες συντάξεις. Πιέτη Κάινεν, Κρόιτσμαν, Τούρινεν από τους Πρασίνους και εγώ είμαι σκιώδης από τους Ευρωπαίους μεταρρυθμιστές και συντηρητικούς. Η κυρία Μάτικ είναι εδώ. Από την Κομισιόν έχουμε κάποιον. η Κομισιόν θα λάβει το, το λόγο επί του θέματος. Όχι, όχι, δεν έχουμε κανέναν από την Κομισιόν. Ωραία, θα δώσω το λόγο στον κύριο Κοφεράτη για να μιλήσουμε για τη τροπολογίες συμβιβασμού. Μετά θα ακούσουμε τους ε, σκιώδεις και αύριο τέλος θα ψηφίσουμε. Κύριε Κοφεράτη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όπως κάνουμε κάθε φορά τελετουργικά, τους σκιώδεις για την εργασία τους και γιατί ήταν ιδιαίτερα διαθέσιμοι στην πιο δεσμευτική φάση όταν αναζητούσαμε τελικούς συμβιβασμούς. Επίσης, οι πολιτικές ομάδες μας στήριξαν και προβλήθηκαν και απαιτήσει οι οποίες επιλήθηκαν στις προτάσεις συμβιβασμού. Οι προτάσεις τους έγιναν αποδεκτές λίγες μέρες πριν. Φτάσαμε σε τροπολογίες συμβιβασμού. Θα ήθελα μόνο να σταθώ εντάχει σε ορισμένα ζητήματα. Το πρώτο, όπως είπαμε και στις ε, προηγούμενες συζητήσεις, και όπως πολύ καλά γνωρίζουν ε, οι σκιώδεις, ένα από τα βασικότερα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν και αυτό είναι θέμα και της Επιτροπής, που είναι ο τελικός αποδέκτης των προτάσεων. Αφορά την δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων και εδώ η Ευρώπη χρειάζεται μεγάλη κινητικότητα γιατί θα προέλθουν και από άλλες ε, χώρες του κόσμου πολίτες οι οποίοι θα εργαστούν για την Ευρώπη και στο τέλος ε, της εργασιακής περίοδου θα πρέπει να ε, κατοχυρωθούν τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα. Αυτό ακριβώς προσπαθήσαμε να καλύψουμε ως προς τη δυνατότητα μεταφοράς στο τέλος μιας δραστηριότητας, μακρόχρονης δραστηριότητας. Γι' αυτό θα πρέπει όλοι να έχουν το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή συνταξιοδότηση. Το θέμα λοιπόν της μεταφοράς είναι ύψης της σημασίας. Γιατί τα μεμονωμένα συστήματα όλο ένα και επικαιροποιούνται έτσι ώστε να έχουμε να κάνουμε με συστήματα επιμερισμού και κεφαλαιοποίησης χωρίς ε, καμία ρήξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα άλλο θέμα το οποίο μας απασχόλησε ιδιαίτερα και όπου υπάρχει σύγκληση απόψεων αφορά τη νέα οργάνωση των συνταξιοδοτικών συστημάτων και των συστημάτων προνοίας, γιατί βασιζόμαστε σε τρία επίπεδα, το δημόσιο σύστημα συνταξιοδοτήσεων, τις επικουρικές συντάξεις ή συμπληρωματικές και για όποιον το επιθυμεί μία επιπρόσθετη ασφάλιση ιδιωτικής φύσης όταν το επιθυμούν οι πολίτες και οι τρεις πυλώνες χρήζουν προστασίας και επικαιροποίησης για να φτάνουμε σε ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα. Γι' αυτό θα πρέπει να οργανώσουμε εκ νέου τους φορείς που ασχολούνται με συστήματα προνοίας και η νέα αυτή οργάνωση θα πρέπει να κινηθεί προς την στοιχειοθέτηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων έτσι ώστε να υπερβούμε τα προσκόμματα τα οποία δυστυχώς υπάρχουν γιατί τα σύνορα πλέον δεν θα πρέπει να μας χωρίζουν όπως έκανε στο παρελθόν. Θα πρέπει να μας οδηγήσουν σε μια γενικότερη ευημερία, σε κράτη προονία, σε welfare states, που είναι πλέον αποτελεσματικά. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα στοιχεία σύγκλησης. Είμαι πεπισμένος και ιδιαίτερα ικανοποιημένος γι' αυτό και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πάντες για τη συνεργασία και ιδιαίτερα τους σκιώδεις με τους οποίους συναντηθήκαμε πολλές φορές. Ωραία, σας ευχαριστώ. Η κυρία Κάινεν. Εγώ από πλευρά μου θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κοφεράτη ιδιαίτερα για την επικοδομητική και θετική δουλειά που έκανε. Όπως επίσης και τις καλές προτάσεις του συμβιβαστικές αλλά και συνολικά. Και θέλω να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους και του εισηγητές για μια πολύ επικοδομητική συνεργασία. Νομίζω ότι καλύψαμε, σημαντικά θέματα. Τη γύρανση του πληθυσμού, τις πιέσεις από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, όπως επίσης και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα διάφορα κράτη-μέλη ε, σε σχέση και με τα δύο φύλλα. Τώρα για τους συμβιβασμούς βρήκαμε πολύ θετικό και ισόρροπο τρόπο να προχωρήσουμε με τη σειρά προτιμήσεων των διαφόρων πεδίων, των διαφόρων πυλώνων, ο δημόσιος πυλώνας ας πούμε και μετά η βελτίωση και η επέκταση τα συμπληρωματικά συνταξιδοτικά προγράμματα, τις επικουρικές συντάξεις και άλλα και να ενθαρρύνουμε τα ιδιωτικά. Είναι πολύ σημαντικό για μας να υπάρξει ένας καλός συμβιβασμός, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να, να ε, συναρτήσουν την, ε, αγορά, την ε, ηλικία συνταξιοδότησης με, το προσδόκιμο ζωής, δηλαδή θα πρέπει να μην είναι υποχρεωτικά, αλλά να υπάρχουν δυνατότητες επιλογών. Τέλος, η δυνατότητα μεταφοράς των συντάξεων. Με τα σχόλια αυτά, με τα χαράς, αποδέχομαι το τα προτινόμενα συμβιβαστικά κείμενα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω εισηγητή και συναδέλφους για την πολύ καλή συμβαστική λύση που έχουμε βρει. Και θα ήθελα πολύ σύντομα να πω ότι ο πρώτος πυλώνας ε, του ε, συνταξιδοτικού συστήματος βρίσκεται σε πίεση, γι' αυτό ε, ε τη σημασία των, δύο άλλων πυλώνων. Επίσης, ε, ε, πρέπει να ρυθμιστεί ο τρίτος πυλώνας έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε σωστές επιπτώσεις στο σύστημα συνταξιοδότησης. Θα πρέπει να προσέχουμε γιατί οι συμβαστικές προτάσεις έχουν δείξει ότι υπάρχει, ε, υπάρχουν κανόνες ε, 2 για τα συστήματα συντάξεων και ε, τα επαγγελματικά ταμεία δεν πρέπει να είναι στην ελεύθερη αγορά. Από την άλλη υπάρχουν σημεία στα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερους κανόνες, ειδικότερα ε, το θέμα της αποδοτικότητας ε, των ε, συντάξεων όποτε υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα των εργαζομένων και αυτό είναι πολύ σημαντικό στην εσωτερική αγορά γιατί έχουμε υψηλό βαθμό ανεργίας στην Ισπανία και θα μπορούσαν οι άνθρωποι αυτοί να δουλέψουν στη Γερμανία αλλά λόγω της γιατί λόγω της δημογραφικής εξέλιξης δεν έχουμε απογόνους. Θα ήταν καλό λοιπόν να υπάρχει κινητικότητα στην Ευρώπη για τους εργαζόμενους και για την απασχόληση, αλλά αυτό ε, θα πρέπει να αποτελεί και κίνητρο για να μπορέσουμε να βρούμε περισσότερες θέσεις εργασίας και να υπάρχει και μια αποδοτικότητα των συντάξεων. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για αυτήν την συμβαστική λύση και νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλό. Ευχαριστούμε. Η κυρία Τούρνεν, ευχαριστώ τον εισηγητή και τους άλλους σκιώδεις. Ε, νομίζω ότι καταφέραμε να καταλήξουμε σε ένα πολύ καλό σημείο για όλους μας. Ε, είχαμε ε, κάποια μικρά προβλήματα με την συμβαστική λύση 3, πρόταση 3, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Πετικάινεν, η οποία ήταν τόσο ανοιχτή, γιατί τώρα θα είναι επιπρόσθετα τα ιδιωτικά ε, συστήματα συνταξιοδότησης. Ε, υπάρχουν τώρα, είναι ε, επικουρικά, αλλά δεν μπορούμε ως κοινωνία να βασίσουμε τα συστήματά μας εκεί. Γι' αυτό ήταν σημαντικό για μας να υπάρχουν σωστές προτεραιότητες μεταξύ των τριών πυλώνων και γι' αυτό υποστηρίζουμε την πρόταση. Ευχαριστούμε λοιπόν γι' αυτό. Τι άλλο να πω τίποτα. Είμαι ευχαριστημένη. Πολύ ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να μιλήσω κι εγώ εκ μέρους της ομάδας μου. Προσωπικά δεν έδωσα μεγάλη προσοχή σε αυτό το θέμα λόγω άλλων πραγμάτων. Ο κύριος Καπεράτη δεν ήταν υπέρ ε, κάποιων των ε, τροπολογιών γιατί ήταν ε, πολύ δύσκολο να γίνουν αποδεκτές όλες αλλά από τη δική μου πλευρά νομίζω ότι ήταν σημαντικό στη γνωμοδότηση να αναφέρεται, να υπάρχει μια γεύση του γεγονότος ότι βασικά είναι ευθύνη του κράτους οι συντάξει. παραμένουν ευθύνη του κράτους και υπάρχει μια συγκεκριμένη τροπολογία όπου εφιστούσα την προσοχή στο γεγονός ότι σύμφωνα με τη μέθοδο που υπάρχει ε, τα κράτη-μέλη έχουν ε, ε, συμφωνήσει να παρακολουθούν κάποιους δείκτες και η Κομισιόν έχει συμφωνήσει να επικεντρωθεί σε αυτό το συμφωνημένο πορτφόλιο, σε αυτό το φάκελο, παρά να προτείνει νέα πράγματα. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν ρεαλιστές. Όσον αφορά στις συμβαστικές τροπολογίες, υπάρχουν πολλές από τις τροπολογίες μας που έχουν συμπεριληφθεί σε αυτές, χωρίς να υπάρχουν πολλές αλλαγές. Ε, νομίζω ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε την συμβαστική ένα, στην οποία δεν θα μπορέσουμε να, να υποστηρίξουμε την ε, τροπολογία 1, τη συμβαστική, γιατί δεν συμπεριλήφθηκαν αυτά που θέλαμε και δεν συμφωνούμε με τη διατύπωση. Είμαστε υπέρ τη αρχικής διατύπωση του κ. Κοφεράτσι. Γενικά νομίζω ότι μπορούμε να συμβάλλουμε στο θέμα της εσωτερικής αγοράς και όπως έχω πει πολλές φορές θέλουμε να έχουμε προστιθέμενη αξία. Έτσι πρέπει να συμβάλλουμε εμείς όπως και η Επιτροπή Απασχόλησης. Πρέπει να δίνουμε στους ε, εργαζομένους ε, τη δυνατότητα μέσα στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς να έχουν προστιθέμενη αξία. Αύριο ε, θα δούμε αν θα δώσουμε την αμέριστη υποστήριξή μας στην έκθεση. Θα συμβουλευτώ πρώτα του συναδέλφου μου. Είναι η πρώτη ή δεύτερη έκθεση του κυρίου Κομφεράτη και πραγματικά φαίνεται ότι έχει αποκτήσει εμπειρία στο να βρίσκει καλούς συμβεβασμούς. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο από την Κομισιόν εδώ, μάλλον όχι. Οπότε καλώ τον κύριο Κοφεράτη να ολοκληρώσει την ε, σημερινή συζήτηση. Η Επιτροπή συνταξιοδοτήθηκε, από ό,τι φαίνεται. Ένα στοιχείο μόνο θα ήθελα να αναφέρω. Συμφωνώ με αυτά που είπατε λίγο πριν. Νομίζω ότι η εργασία μας θα πρέπει να επικεντρώνεται σε τέτοια θέματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε πραγματικά να προβάλλουμε μια πραγματική προστιθέμενη αξία υπέρ των ε, πολιτών. Το θέμα της δυνατότητας μεταφοράς είναι ύψης της σημασίας για, τις για τους πολίτες μας και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να το προωθήσουμε. Εγώ συμμετείχα στην Πράσινη Βίβλο για τα συνταξιοδοτικά, για το συνταξιοδοτικό και εδώ επικεντρώνεται η Επιτροπή σε θέματα δικαιωμάτων. Θα πρέπει όμως να νομοθετήσουν τα κράτη-μέλη όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλά να προσδώσουμε κοινωνική, κοινοτική με συγχωρείτε, διάσταση σε ορισμένα θέματα ως προς τη μεταφορά δικαιωμάτων και το περιεχόμενο του πλαισίου πρόνοιας. Είναι ένα θέμα εσωτερικής αγοράς και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει αποτελεσματικά να βοηθήσουμε την Επιτροπή Εργασίας. Διαφορετικά, δεν θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε θέματα ουσίας μέσα στα πλαίσια της Ένωσης στην οποία κινούμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Θα ψηφίσουμε αύριο και για αυτή την έκθεση. Άρα ολοκληρώνουμε τις σημερινές εργασίες γιατί όπως σας είπα σήμερα δεν θα γνωμοδοτήσουμε επί της έκθεσης Τρατσκόφσκι γιατί δεν είχαμε όλες τις τροπολογίες, δεν είχαν μεταφραστεί όλες οι τροπολογίες. Θα συναντηθούμε αύριο το πρωί στις 9 για να ασχοληθούμε με τις τροπολογίες μέσα στα πλαίσια της ευθυγράμμισης ε, σε επίπεδο επιτροπολογίας για τα αγαθά. Μετά ο κύριος Αρίας θα μας πει τι γίνεται με το ηλεκτρονικό ε, εμπόριο και θα αρχίσουμε την ψηφοφορία στις 10. Ε, Έχουμε 600, α, 900 τροπολογίες μου υπενθυμίζει η γραμματεία σε δύο ώρες που πρέπει να ψηφίσουμε. Ελπίζω να τα καταφέρουμε με όλους τους συμβιβασμούς. Στις 10 όλα αυτά. Μετά έχουμε τη δεύτερη γνωμοδότηση κοφεράτη στις 12. Και το απόγευμα έχουμε την ε, παρουσίαση της Κυπριακής Προεδρίας το θέμα του προϋπολογισμού. Άρα έχουμε μία ε, μεγάλη ημέρα εργασιών πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Σας ευχαριστώ πολύ και θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9.